Dear colleagues, we can start our meeting. Αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας, κυρίες και κύριε, Κύριε, είναι εδώ η Ιαν Κέλερμαν, η Τζόαν Κέλερμαν για επίσημη ακρόαση από τότε που η Επιτροπή την όρισε υποψήφια για τη θέση του μέλους του Συμβουλίου του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγένσης. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια βεβαίως. Ε, γνωρίζετε ότι μέλη της ε, ομάδας της Τραπεζικής Ένωσης και άλλα ε, μέλη είχαν ήδη ανταλλαγή απόψεων και κλεισμένων των θυρών με την κυρία Κέλερμαν και με άλλους επιλεγέντες υποψηφίους στο πλαίσιο μιας θετικής και επικοδομητικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του Συμβουλίου. Τώρα έχουμε φτάσει στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αυτής που είναι η επίσημη ακρόαση της κυρίας Κέλερμαν η οποία είναι εκτελεστική διευθύντρια και ε, μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολλανδικής ε, Κεντρικής Τράπεζας και θα ήθελα να της δώσω τώρα το λόγο για να μας κάνει εισαγωγικά σχόλια 5 λεπτών κατόπιν των οποίων θα γίνει ένας γύρος ερωταποκρίσεων. Κυρία Κέλερμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, βουλευτές μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας ε, και για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Είναι τιμή και προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης που είναι το, ε, συμβούλιο, το ενιαίο Συμβούλιο εξηγένση, αν δούμε του δύο πυλώνε που υφίστανται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας ως ε, ένα ε, ως ε, γενικοί παθολόγοι και νοσοκόμοι που προσπαθούν να κρατήσουν τον τραπεζικό τομέα υγιή και να τον φροντίσουν. Αν δει κανείς όμως το SRB, ε, το Συμβούλιο δηλαδή, είναι τα κατεπήγοντα. Είναι τα επίγοντα περιστατικά ε, στα οποία δεν θέλουμε να πάει κανείς. Αν όμως χρειάζεται κάποια τράπεζα να πάει στα επίγοντα, πρέπει να είναι έτοιμα τα επίγοντα να την υποδεχθούν. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτό το σημαντικό καθήκον. Ο λόγο είναι ότι έχουν, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Πριν από την οικονομική κρίση είχαμε αρχίσει να βλέπουμε ότι υπήρχε το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο ε, και είδαμε ότι υπήρχαν πολλέ τράπεζε που εκμεταλλεύονταν αυτέ τι δυνατότητε και ήταν πολύ ενεργοί εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό αυτή. Παρ' αυτά δεν υπήρχε καμία εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η αρχή ε, καν της εξυγίανσης δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν κανόνες, δεν υπήρχαν ε, εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και ξαφνικά ήρθε η ε, κρίση με την κατάρρευση της Lehman Brothers, κάτι το οποίο συγκλώνησε την Ευρώπη και εγώ συμμετείχα προσωπικά σε δύο προσπάθειες με τις ε, Ολλανδικές αρχές και τις Βελγικές αρχές και τις αρχές της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου για να σώσουμε ε, μια ανοιχτή τη φόρτης την τράπεζα φόρτης και προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά μια τρομακτική εμπειρία για την ώρα έχουμε καταφέρει να τη σώσουμε από πλήρη κατάρρευση. Για μένα όμως απέστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ε, η διαδικασία, η κατάσταση αυτή είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ξανασυμβεί. Και τώρα έχουμε τους κανόνες και τα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τραπεζών που είναι πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν και έχουμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε μια απειλή στους φορολογούμενους. Για μένα θα ήταν λοιπόν ένα προνόμιο να συμμετέχω σε αυτήν σε αυτό το ε, εγχείρημα. Έχω εμπειρία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρω ε, πόσο περίπλοκο είναι να γίνει κανείς ε, μια μεγάλη διασυνοριακή συναλλαγή με πολλά μέρη που συμμετέχουν, με τράπεζες που είναι πολύ δραστήριες στην αγορά κεφαλαίων, με το κυβερνητικό πλαίσιο και τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Αλλά πιστεύω ότι το, συμβούλιο, το ενιαίο Συμβούλιο εξηγεί Intelligences μπορεί πράγματι να ε, βοηθήσει. Ο προγραμματισμός εξυγίανσης είναι το πιο σημαντικό. Να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι πάρα πολύ περίπλοκες ούτε πολύ μεγάλες οι τράπεζες για να πτωχεύσουν και να μπορούν να εξυγιανθούν ε, με, τα, ε, με σωστό τρόπο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν το Συμβούλιο να κάνει κάτι τέτοιο, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να σταματήσουν τη λειτουργία τους οι τράπεζες με σωστό τρόπο, όχι και άτακτα, με, χωρίς ε, επιπλέον βάρος ούτε για το πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ούτε για τους φορολογουμένους. Για, ε, ε, τι πρέπει να κάνει το Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρόβλεψη, η πρόληψη, ο προγραμματισμός της εξυγίανσης, αλλά και η αποφυγή της εξυγίανσης. Αν όμως φτάσει το πράγμα σε εξυγίανση, τότε το Συμβούλιο ε, αυτό πρέπει να έχει μια ουδέτερη στάση, να είναι ανοιχτό και διαφανές και στα ε, μέλη ε, και εκτός των μελών της Ευρωζώνης, γιατί δεν είναι όλες οι τράπεζες οι ίδιες, ούτε όλες οι καταστάσεις ίδιες. Θα πρέπει να γίνει εξισορρόπηση του συμφέροντος της ε, ανησυχίας ε, για τις τράπεζες αυτές, αλλά ε, και τη σταθερότητα της οικονομίας. Αν λοιπόν επιλεγώ, ποιο θα είναι το όραμά μου για το Συμβούλιο αυτό. Καταρχάς, είναι μια αρχή που πρέπει να λειτουργεί σε ένα πολύ περίπλοκο πεδίο με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο θα είμαστε υπόλογοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικές Αρχές Εξυγίανσης, ο ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης, οι τράπεζες, οι ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε στενά, αλλά θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη αυτή η αρχή. Επίσης, ε, θα χρειαστεί να γίνει πολλή δουλειά, αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε αυτή ε, η δουλειά θα χρειαστεί να γίνει από το Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι και να ε, προσπαθήσουμε να προλάβουμε καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε και αξιόπιστοι. Πρέπει το Συμβούλιο να μπορεί να δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση και να δείξει ότι θα χρειαστεί το bail-in, ε, αν χρειαστεί, θα χρειαστεί να είναι πολύ καλή επικοινωνία, να διαχειριστεί ε, σωστά την κρίση με έναν αξιόπιστο, και, ε, με έναν αξιόπιστο τρόπο και ε, με λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very... Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον πρωτομιλητή, κ. Ζάλμπα από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε, αγαπητή υποψήφια. Έχω μία ερώτηση να σας θέσω, μία συγκεκριμένη ερώτηση. Σε περιπτώσεις εξηγίανσης που περιλαμβάνουν και κρατικούς πόρους, τι μέτρα θα λάβατε για να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των αποφάσεων του SRM και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή που μου θέσατε. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό το οποίο αναφέρετε. Νομίζω ότι η προκαταρτική απάντηση είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κρατικές ε, ενισχύσεις, επιδοτήσεις του τουλεχθέντος, να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο ζητημάτων. Είναι μια πολύ ε, λεπτή ισορροπία με το κανόνον, στον κανονισμό για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι υπάρχει ένα σύστημα σωστής συμμετοχής για το ενδεχόμενο και την ενδεχόμενη κριτική ενίσχυση. Αλλά υπάρχει και μία άτυπη οδός. Θα πρέπει να υπάρχουν και ανεπίσημες ε, επαφές και επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει παρανόηση. Αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο. Αν χρειαστεί να επισέλθουμε στην διαδικασία λήψης απόφασης του άρθρου 18 θα πρέπει να γνωρίζουμε το τι συζητάμε, να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Υπάρχει λοιπόν ένας ε, επίσημος, τυπικός τρόπος επικοινωνίας, αλλά θεωρώ ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος επικοινωνίας ε, άτυπα, ανεπίσημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν ε, θέλετε να κάνετε κάποια επερώτηση, έχετε πέντε λεπτά συνολικά στη διάθεσή σας. Ο κ. Μπαϊέ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε η Τρία Σερμαν που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική η ευθύνη του Συμβουλίου γιατί αποτελεί και πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση. Εμείς οι σοσιαλιστές ε, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση ε, σε αυτό το ζήτημα, ώστε να μην έχουμε και πάλι φαινόμενα όπως η κρίση του 2008. Γιατί είδαμε την κοινωνική τραγωδία που προκλήθηκε ε, στην, και στον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη και κάτι το οποίο τονίστηκε ιδιαίτερα και χθε στην απεργία εδώ στο Βέλγιο. Τα stress test έχουν ήδη δείξει ε, προβλήματα σε, κάποιες, σε κάποια τραπεζικά ιδρύματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιο είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα σας για τα επόμενα χρόνια και ποια είναι τα μέτρα που θα πάρετε για να καταστεί λειτουργικό ώστε να τον πιο γρήγορα ο μηχανισμό για να αποφύγουμε προ όφελο των Ευρωπαίων συμπολιτών μα μία πιθανή τραπεζική πτώχευση. Ευχαριστώ. Thank you. I... Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα αγγλικά. Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει ένα στενόχρονο διάγραμμα για την ε, θέσπιση του Ταμείου. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευθεί. Το πρώτο έτος λειτουργίας ε, του Συμβουλίου Εξεγένσης θα είναι και πολύ σημαντικό έτος. Είναι έτος προετοιμασίας κατά το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός και τα σχέδια εξυγίανσης για τις τράπεζες θα πρέπει να έχουν ε, εκπονηθεί. Πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη χρονιά μια πραγματική, πραγματικά μεταβατική χρονιά. Γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα γιατί το ε, Συμβούλιο θα τεθεί σε ισχύ από το 2016 και μετά. Η προετοιμασία λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Μεγάλο τμήμα της χρονιάς θα το αφιερώσουμε σε αυτό. Όπως ξέρετε, ελπίζουμε σύντομα, ακόμα και σήμερα, <laughs> να ληφθεί απόφαση, να υπάρξει λευκός καπνός, ακριβώς για την ε, σύνθεση του Συμβουλίου γιατί βέβαια αν δεν επιληθεί αυτό δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά. Αλλά όπως είπα ο σχεδιασμός εξηγήσεις είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να διαμορφώσουμε και στενές επαφές με ε, το μηχανισμό εποπτείας, να εξετάσουμε τα αποτελέσματα των stress test και ε, να παρακολουθούμε τις τράπεζες που δεν πέρασαν τα stress test ή τα πέρασαν με δυσκολία για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε αρνητικές και λυσάρε εκπλήξεις το 2016. Σημαντικός είναι και ο ρόλος ε, του μηχανισμού εποπτείας, του SSM, που έχει την εξουσία να προχωρά σε μέτρα ε, πρώιμης παρέμβασης. Είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε και, στην, και στο επόμενο έτος. Αν υπάρξουν τράπεζες που θα πρέπει να υπάρξει τέτοια πρώιμη παρέμβαση, μπορεί να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο αυτές οι τράπεζες να καταλήξουν ε, στα χέρια μας στο Ταμείο Εξυγίανσης. Προετοιμασία λοιπόν, σχεδιασμός εξυγίανσης, προκατακτικές εργασίες, να είναι έτοιμο το Συμβούλιο, αλλά και να αντιλήσουμε διδάγματα από άλλους θεσμούς, οργανισμούς και ιδρύματα, και εδώ αλλά και σε άλλα τμήματα της εφηλίου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά για μας. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, Στάνισλαφ ο Τζοκ από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. τιμή, κυρία Κέλλερμαν. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε εν συντομία ποια είναι η σύνδεση θεωρείται μεταξύ των ε, τραπεζών που βρίσκονται στη διαδικασία πτώχευσης και του μηχανισμού σε ό,τι αφορά και τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι γίνεται, ποια είναι η νομοθεσία και πώς διέπει το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Yes, thank you. Um, you are... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάτε ποια είναι η σχέση μεταξύ της πτώχευσης των τραπεζών και της πρότασης ε, για τη μεταρρύθμιση των τραπεζικού συστήματων σε μία σύνδεση μεταξύ των δύο. Γιατί και οι δύο ομάδες κανόνων έχουν σκοπό να αποτρέψουν την πτώχευση πολύ μεγάλων τραπεζών που είναι πάρα πολύ σύνθετο να πτωχεύσουν. Θεωρώ ότι η σημασία της πρότασης είναι έγκυται στο ότι μας δίνει μέσα για να μειώσουμε την περιπλοκότητα και την ε, πολυμορφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε πολλές από τις τράπεζες. Και το Συμβούλιο Εξυγίανσης ε, θα λαμβάνει υπόψη αυτά. Γιατί θεωρούμε ότι κάποια είδη συναλλαγών όπως ε, τα προβληματικά στοιχεία θα πρέπει να αλλάξουν. Φυσικά υπάρχει σύνδεσμος λοιπόν, υπάρχει διαφορά σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή των ε, μέσων. Η Ευρωζώνη, το σύνολο της Ένωσης, αντίστοιχα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποια άλλη ο στόχος είναι ο ίδιος. Δεν χρειάζονται άλλη επικαλύψεις, θεωρώ. Είναι απαραίτητο οι επόπτες και η ενιαρχή αρχή θα έχουν την αρμοδιότητα να μειώσουν την περιπλοκότητα σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι είναι απαραίτητο αυτό για τις διαδικασίες εξυγίανσης. Yes, for the other group, Mr. Από πλευρά άλλο το κύριο Στόιρερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κέρμα, μία ερώτηση έχω να σας κάνω. Θα μπορούσατε από την επαγγελματική σας εμπειρία ως τώρα να μας αναφέρετε ένα παράδειγμα όπου ήσασταν υπεύθυνοι για διαχείριση κρίσεων γιατί με τη νέα σας αρμοδιότητα θα αναγκαστείτε ουσιαστικά αυτό να κάνετε, διαχείριση κρίσεων. Στην επαγγελματική σας εμπειρία λοιπόν υπάρχει ένα παράδειγμα που μπορείτε να καταδείξετε πώς αντιδράσατε για να μας δείξετε ποια είναι η εμπειρία η οποία, την οποία έχετε. Η απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και ασφαλώς είναι πολύ έγκυρο και εύστοχο το ερώτημα αυτό προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το SRB θα είναι ε, έτοιμο για διαχείριση κρίσεων Έχω επαγγελματικό υπόβαθρο ως δικηγόρος και αυτό μου δίνει μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά την ανάλυση συναλλαγών ε, κεφαλαγορών. Δεν ήταν μεν διαχείριση κρίσεων, αλλά μου έχει δώσει σημαντική εμπειρία της έκθεσης στις κεφαλαγορές αργότερα. Όταν ε, έγινα διευθύντρια στην, Ευρωπαϊκή, στην Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, Δυστυχώ αναγκάστηκα να έχω πιο πολλή εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων από ό,τι θα ήθελα και από ό,τι θα πίστευε κανεί. Ξεκίνησαν τα πράγματα με την οικονομική κρίση. Εγώ ξεκίνησα, ξέρετε, στα τέλη του 2007. Και τότε λοιπόν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της κρίσης. Ε, συμμετείχα στην διαχείριση της κρίσης της Φόρτης, το οποίο φυσικά ήταν μια διασυνοριακή υπόθεση αλλά εκ παραλλήλου στην Ολλανδία είχαμε το iSafe, την ING, την τράπεζα, η οποία επίσης ε, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και χρειάστηκε κρατητική επιδότηση. Είχαμε την Eichol, είχαμε την τράπεζα SNS Real και πολύ φοβάμαι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η συμμετοχή η προσωπική μου ήταν μεγάλη. Μεγάλη μερίδιο λοιπόν συμμετοχής και πρόσφατα αναγκαστήκαμε να ξαναεπανέλθουμε στο θέμα της SNS Real, μια, μια εταιρεία η οποία ιδιωτικο... Ε, αναλήφθηκε από το Ολλανδικό Δημόσιο το 2014 και έγινε ένα είδος bail-in. Συμμετείχα λοιπόν στις περισσότερες κρίσεις που εμφανίστηκαν στην Ολλανδία και νομίζω ότι αυτό μου έδωσε μια εμπειρία που θεωρώ ότι θα είναι πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη σε περίπτωση που επιβεβαιωθώ στη θέση αυτή. Sven Giegold. Σβέν Sven Giegold. Sorry. είχα ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή μου. Ένα ερώτημα. Είστε από τις κατοχώρες σας. Στην νομοθετική βάση είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για πιθανές τρευλώσεις ε, όταν συγκρίνουμε ένα εθνικό σύστημα τραπεζικής εξυγίανσης και χρηματοδότησής του και αφετέρου ένα ευρωπαϊκό τέτοιο σύστημα. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια στρέβλωση ότι δηλαδή σε ένα ε, εθνικό σύστημα με υψηλή συγκέντρωση, ε, με χαμηλές ε, σταθερέ καταθέσεις, ότι αυτές οι τράπεζες θα χρειαστούν να πληρώσουν περισσότερα σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα από ότι σε ένα καθαρά εθνικό. Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί στρέβλωση ότι δηλαδή αυτές οι τράπεζες θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα από ότι σε ένα εθνικό. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα έχει αρμοδιότητες για να εξετάσει ακριβώς και αυτό το ζήτημα της κατανομής. Κυρία Κέλλαρμαν, ευχαριστώ. Εξαιρετικά επίκαιρο το ερώτημα. Ομολογώ ότι δεν ξέρω τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά αυτές τις συζητήσεις. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας δώσω μια γενική απάντηση. Να μην υπησέλθω ε, σε συγκεκριμένο παράδειγμα χώρας. Εν γέννη, είναι καλό οι τράπεζες που παρουσιάζουν και να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πληρώνουν περισσότερο. Είναι μια γενική αρχή αυτή που έχει, που έχει υιοθετηθεί. Και νομίζω ότι ορθώς υιοθετήθηκε. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σας πω έτσι αυτή τη στιγμή απ' έξω τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Είναι πάντα ιδιαίτερα περίπλοκη αυτή η συζήτηση. Και από την εμπειρία μου στην προηγούμενη μου θέση είδα ότι είναι δύσκολο να το προσδιορίσει κάποιο αυτό. Γιατί πάντα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, αλλά, ναι, αλλά σε σχέση με τι. Επομένω, η στάθμιση κινδύνου είναι κάτι θετικό με την ε, ενίδια συμφορών, συγγνώμη, εισφορών, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι ε, ακριβώς από εκεί πέρα. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το ζήτημα. Επερώτηση. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε εδώ που έχουμε συνήθω, αλλά είναι πολύ απλή η παρατηρήσή μου. Αν βασιζόμαστε σε καταθέσεις, τουλάχιστον υπάρχει μια σχετική σταθερότητα σε σχέση με κάποιον ε, που πηγαίνει σε ε, πλήρη χρηματοδότηση. Και αυτή είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή μεταξύ κρατών μελών και συμβουλίου, όπου με βάση και τους πίνακες που έχουμε λάβει, η κατανομή υπολογίζεται όχι βάσει κράτους μέλους και όχι βάση της τράπεζας και του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτή είναι η συζήτηση που εμένα με ενδιαφέρει. Το ζήτημα κατανομής μεταξύ κρατών μελών από πλευράς μου δεν αποτελεί στρέβλωση. Το Συμβούλιο διαστρεβλώνει το πνεύμα του κανονισμού και είναι ιδιαίτερα παράξενο αυτό κατά τη γνώμη μου αλλά μπορείτε αυτό να το λάβετε ως ε, σχόλιο. Ναι, ως σχόλιο θα το λάβω. Λέει η κυρία Κελέρμαν, μία μόνο παρατήρηση εν είδη απάντησης. Κατανοώ αυτό που λέτε, όμως παραμένει εξαιρετικά δύσκολο το ζήτημα, γιατί έχουμε δύο πυλώνες στην Τραπεζική Ένωση, όμως δεν έχουμε Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Εσείς μιλήσατε για καταθέσεις. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλη διαφορά ο τρόπος διασφάλισης τους και πώς ακριβώς αυτό θα λειτουργήσει. Θα παραμείνει λοιπόν αυτό το ζήτημα, πιστεύω, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Μόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, ε, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Κέλλερμαν Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω που συχνά ανακύπτει στο μυαλό μου Συνεχώς μας ανακοινώνεται ότι περισσότερο χρησιμοποιείται το bail-in αντί το bail-out για να μην χρειάζεται να πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Είδαμε όμως ε, τη σύνθεση των τραπεζών ε, και των καταθέσεων, κυρίως ιδιώτες είναι αυτοί και συνήθως είναι φορολογούμενοι αυτοί οι καταθέτες. Οπότε οι φορολογούμενοι και οι πελάτες των τραπεζών ε, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί λοιπόν συνεχώς προσπαθείτε να αποφύγετε την επανεθνικοποίηση στην περίπτωση ενός συστημικού κινδύνου που έχει εμφανιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και νομίζω ότι αναφέρεστε σε ένα σημαντικό θέμα που είναι το εξής. Πώς ακριβώς δουλεύει το bail η διάσωση με ίδια μέσα σε σχέση με την διάσωση την απλή και πώς είναι δυνατή, δυνατό να προστατεύσει κανείς και τους καταθέτες και τους φορολογουμένους. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του κανονισμού και ο σκοπός ολόκληρου του συστήματος. Νομίζω ότι για κάθε σύστημα προκειμένου να λειτουργήσει είναι σημαντικό οι κανόνες του παιχνιδιού να είναι σαφέστατοι από την αρχή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό καθήκον ε, για το ε, Συμβούλιο Εξυγίανσης ε, πριν αρχίσουν να ισχύουν οι κανόνες για το Μπέιλιν το 2016 να εξασφαλίσουμε το τι σημαίνει και το τι δεν σημαίνει τι ακριβώς θα, ποιοι ακριβώς θα έπρεπε να γνωρίζουν τις πιθανότητες Μπέιλιν και ποια είναι η θέση των επενδυτών που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο του Μπέιλιν και να ξέρουν τι να περιμένουν, να μην εκπλαγούν, γιατί κατά την άποψή μου Υπάρχουν προβλήματα όταν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα προσπαθήσει πάρα πολύ να καταλάβει ποιος είναι, ποια είναι η φύση των κανόνων για τον Μπέιλιν και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των κανόνων αυτών. Αυτό είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του ρόλου μας, γιατί όταν υπάρχει τράπεζα που αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι πολύ αργά να αρχίσουμε τότε να επικοινωνούμε για τέτοιου είδους ζητήματα. Πρέπει να είμαστε σαφείς και στους ε, καταθέτες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και γνωρίζουν σε ποιο βαθμό ε, υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε bail Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, το κλειδί βρίσκεται στην προετοιμασία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το bail όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Βαντεν Κελάρτε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την καλή σα προφορά. Κυρία Κέλερμαν, ε, μία βελγική ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σα ε, για την παρέμβαση ε, του Συμβουλίου σε σχέση με τα μοντέλα, για παράδειγμα, ασφαλίσεων υπάρχει περίπτωση εποπτείας κατά τη διάρκεια κρίσης ή ένα τέτοιο μοντέλο όπως και ένα επιχειρηματικό μοντέλο θα έπρεπε να υποφελείται από ε, ένα μοντέλο διαφοροποίησης των κινδύνων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κέλερμαν. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα αυτό και είναι πολυ λεει η κυρια κελλερμαν ειναι ενα πολυ καλο ερωτημα αυτο και ειναι κατι το οποίο το έχω σκεφτεί πολλές φορές και στη δική μου χώρα γιατί το ε, μοντέλο τραπεζικών ασφαλίσεων ε, ήταν κυρίαρχο και στη δική μου χώρα. Φοβούμαι ότι η ερώτησή σας είναι πολύ περίπλοκη για να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι. Υποθέτω ότι αυτό θα περιμένατε. Η πραγματική απάντηση όμως είναι εξαρτάται. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε πολύ καλά το επιχειρηματικό μοντέλο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι από την επόμενη χρονιά θα έχουμε για ασφάλεια το Solvency το 2 ε, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο διαφανή σε σχέση με το τι γίνεται στον τομέα των τραπεζικών ασφαλίσεων και πώς, πώς μπορεί να γίνει η εξισορρόπηση των κινδύνεων πόσο, σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί να γίνει αυτή η εξισορρόπηση κινδύνων. Τούτου λεχθέντος βέβαια στον τομέα των ασφαλίσεων υπάρχει ε, είναι λιγότερο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι θα ήταν στον υπόλοιπο τραπεζικό τομέα και για μένα αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα το μοντέλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να εξετάσουμε προσεκτικότερα και να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην λειτουργεί. Οι Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Υποψήφια, μία ερώτηση που συνεχίζει την προηγούμενη ερώτηση. Πάντοτε αποτελούσε πεποίθησή μου ε, όταν άρχισε να κερδίζει έδαφος η Τραπεζική Ένωση ότι αυτό θα είχε αντίκτυπο για τον τομέα των ασφαλίσεων. Μιλήσατε για το θέμα αυτό συγκεκριμένα, αλλά γενικά όταν γίνεται ανάλυση κινδύνου, μήπως θα έπρεπε κάποια δεδομένη στοιχεία να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο ερώτημα, με την Τραπεζική Ένωση και προφανώς μπαίνετε σε ένα από τα όργανα αυτής της Τραπεζικής Ένωσης. Από τη μία έχουμε μια πολύ ομοσπονδική προσέγγιση κοινοτική ολοκλήρωσης, πολύ ισχυρής με τον μηχανισμό εποπτείας και όταν φτάσαμε στο θέμα της εξυγίανσης ε, επιστρέψαμε σε μια πολύ κυβερνητική μέθοδο που ο καθένας υποστήριξε τη δική του εθνική ε, μέθοδο ίσως θα έπρεπε, είπατε κι εσείς ότι η αξιολόγηση κινδύνου, εντάξει δεν υπάρχει κανένα μαγικό χάπι για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ένα κίνδυνο. Μήπως λοιπόν θα ήταν καλύτερο να ε, βρούμε ένα σύστημα πιο κοινοτικό, να υπάρξει ένα σύστημα ε, φορολόγησης των τραπεζών, κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε το Ταμείο Εξυγίανσης. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δύο είναι οι ερωτήσεις από ό,τι κατάλαβα. Το πρώτο θέμα αφορά τις ε, ασφάλειες. Ε, με ρωτήσατε μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε, όπως έχουμε και τραπεζική ένωση, να έχουμε και μία ένωση ε, ασφαλίσεων. Μπορεί να είναι καλή ιδέα αυτή, αλλά επειδή εγώ έχω αναμειχθεί στην εποπτεία ε, και των τραπεζών και των ασφαλίσεων, πρέπει να πω ότι το πλαίσιο εποπτείας για τις ασφαλίσεις ήταν πραγματικά ε, σε κατάσταση που χρειαζόταν επιγόντως ε, μια διαχείριση και είναι καλό το ότι επιτέλους μπορούμε να το κάνουμε αυτό τον εφαρμόσουμε όμως το μοντέλο που θέλουμε εποπτείας Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι να χωνέψει το σύστημα τις ιδέες του Solvency 2 και να είναι πιο όριμο για το επόμενο στάδιο. Θα μπορούσα βέβαια να φανταστώ ότι κάποια στιγμή ναι, θα κινηθούμε και προς μια ένωση ασφαλίσεων, όπως κινηθήκαμε και προς μια ε, τραπεζική ένωση. Βέβαια δεν είναι τραπεζικά προϊόντα οι ασφάλειες, οπότε ίσως ε, θα έπρεπε να υπάρξει κοινοτική ολοκλήρωση και σε άλλους τομείς, όπως τη φορολόγηση και σε άλλους τομείς, για να υπάρχει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό ε, προϊόν ασφαλίσεων. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε λίγο περισσότερη δουλειά σε αυτό το τομέα από ό,τι έχουμε στον τραπεζικό τομέα. Τώρα, για το γεγονός ε, του Ταμείου και για το γεγονός ότι υπήρχε συζήτηση του κατά πόσο κοινοτικό ή πόσο διακυβερνητικό θα έπρεπε να είναι, νομίζω... Κοιτάξτε, είμαι ρεαλίστρια και σήμερα βλέπω μπροστά μου έναν κανονισμό που υπάρχει δεν θα μπορούσα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα να φανταστώ ότι θα προχωρούσαμε τόσο πολύ σε τόσο μικρό διάστημα στον τομέα της Τραπεζικής Ένωσης. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό επίτευγμα όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ότι έχουμε φτάσει τόσο μακριά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε φτάσει ως εδώ. Νομίζω ότι είναι ένας ε, ε, τρόπος ε, να προχωρήσουμε πολύ βιώσιμος και πραγματικά αναμένω εναγωνίως να αρχίσουμε τη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κέλλερμαν, σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση, πολύ θετική. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή την επόμενη Δευτέρα και αμέσως ε, μετά στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας. colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντόμινικ Λάμπολιο. Αναπληρωτή γενική, Γενικό Γραμματέα Επικεφαλής της ε, Γαλλικής Αρχής ε, Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην Επιτροπή μας για την επίσημη ακρόαση μετά την επίσημη πρότασή σας από την Επιτροπή ως υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή στον, ε, στον Ιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Μετά την ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων διοργανώνεται και η επίσημη ακρόαση και όπως ξέρουν οι συνάδελφοι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαμπολιό για την ε, συνεργασία του με την Επιτροπή μας. Και θα θέλαμε να σας δώσουμε το λόγο για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη, για τη φωνή μου σήμερα. Ελπίζω να είμαι κατανοητός. Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα, κυρίε και κύριοι. Γνωρίζω την Επιτροπή σας και ξέρω ότι και η Επιτροπή σας και το Κοινοβουλίο έχει εμπλακεί και έχει συμμετάσχει έντονα στην αναδιαμόρφωση του συστήματος για την ανταπόκριση στην κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν που βρίσκομαι εδώ σήμερα στον πυρήνα αυτού του σώματος ε, που έχει αντιδράσει στις κρίσεις. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ποιος είμαι και ποιο είναι το έργο μου. Για μένα το Συμβούλιο Εξυγίανσης αποτελεί ένα σύστημα, ένα σαφές συστατικό της ε, Τραπεζικής Ένωσης και είναι σημαντικό λοιπόν, θα είναι μεγάλη μου τιμή να διαδραματίσω ρόλο ρόλος αυτό το νέο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ιστορίας σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα. Είναι σημαντικό αυτό για μένα, γιατί σαφώς θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις στην κρίση. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες άλλωστε. Και τώρα... Εσείς μας έχετε δώσει το σκέλετο και εμείς θα πρέπει να τον ντύσουμε πλέον για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτές των πολιτών, των κρατών και πολλών άλλων εμπλεκομένων φορέων. Τέλος την κρίση, τέλος τον οικονομική και κοινωνική, στο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Σε αυτά που ζήσαμε το 2008. Είμαι πολύ πρόθυμος να διδραματίσω το ρόλο μου και θα κάνω ό,τι μπορώ ως επικεφαλής της σχετικής γενικής διεύθυνσης στη Γαλλία σήμερα κατανοώ τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από τις τράπεζες προκειμένου να σταθεροποιηθούν περισσότερο και να είναι πιο ανθεκτικές αλλά και τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλουν και οι αρχές, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης, αλλά και αυτή η νέα αρχή, αυτό το νέο Συμβούλιο Εξυγίανσης σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ενιαία Εποπτική Αρχή στη Φραγκφούρτη και τις εθνικές ε, αρχές και όλα τα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το καθεξής. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και μάλιστα χρειαζόμαστε μη συνεργασία σε ένα σαφές πλαίσιο, με ένα σαφή συντονισμό. Προετοιμασία και συντονισμό λοιπόν χρειαζόμαστε. Αυτά είναι τα δύο κλειδιά προετοιμασίας για τις κρίσεις. Και θα πρέπει να ενταχθούν αυτά στο σωστό θεσμικό πλαίσιο. Αν θέλουμε να απαντήσουμε στην σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του νέου αυτού σώματος και των άλλων σωμάτων, θα πρέπει να δώσουμε γρήγορες απαντήσεις φτιάχνοντας ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΚΤ, με τις άλλες ε, θεσμικές μονάδες και με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται στον τραπεζικό τομέα. Είναι μεγάλη πρόκληση, το γνωρίζω αυτό. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι εγώ θέλω να παίξω ρόλο στη διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να είμαι διευθυντή ε, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό εξυγίανση, γιατί με ενδιαφέρουν οι συγκεκριμένε δράσει για, το κάθε θεσμικό όργανο. Η συνεργασία, η εξυγίανση για όλους, αλλά και για τις πιο συστημικές τράπεζες σε όλο το παγκόσμιο προσκήνιο, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή ευρωζώνη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ό,τι αφορά και τις τρίτες χώρες. Και ξέρω ότι το να είμαι μέλος του Συμβουλίου σημαίνει μια μεγάλη ευθύνη, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, έχοντας εμπειρία από διάφορα είδη κρίσεων. Είναι σαφές λοιπόν για μένα ότι πρόκειται για ένα εργαλείο κλειδί με σημαντικές ε, ευθύνες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα εξυπηρετήσω το κοινό συμφέρον και ότι θα είμαι υπόλογο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ο σκοπός όλων των κανόνων για το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι το να προληφθούν οι δημόσιες επιδοτήσεις, οι κρατικές ενισχύσεις, αλλά και ο οικονομικός και κοινωνικός αντικτύπος για όλους στην Ευρώπη. Αυτή είναι η στόχη που έχουμε θέσει. Και νομίζω ότι μπορούμε να τους επιδιώξουμε. Και καταρχάς θα πρέπει να είμαστε διαφανείς για να δικαιολογήσουμε, να νομιμοποιήσουμε τις δράσεις μας. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ σήμερα έχω να επιδείξω κάθε δέσμευση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο. Θα κάνω την περνάει από το χέρι μου για την επιτυχία της νέας αυτής, του νέου αυτού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι θα είμαι σε εσάς και προφανώς θα δράσω αμερόλεπτα και ανεξάρτητα, τίμια, έντιμα και ειλικρινά, πέρα από κάθε προσωπικό συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτος ομιλητής, ο Παύλος Ζαλμπά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένα σημείο προγραμματισμού μόνο. Σε περίπτωση έλλειψης ε, μηχανισμών ε, στήριξης ε, και ανάσχεσης. Έχετε κάποια μέτρα ε, που θα προτείνετε να ληφθούν σε περίπτωση που υπάρξουν ανάγκες ε, ανακεφαλαιοποίησης. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Η οδηγία BRRD και ο κανονισμός βασίζονται στην ιδέα ότι θα υπάρχει, ή μάλλον ότι δεν θα χρειαστεί πλέον ένα σύστημα δημόσιας στήριξης. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε το Ταμείο Εξυγίανσης, να, πρέπει να οργανώσουμε ένα προηγούμενο bail-in κάποιων ε, ε, παθητικών και υποχρεώσεων στον ισολογισμό. Ξεκινώντας από τα πιο βασικά, και με το bail-in γίνεται, γίνεται bail-in μάλλον 8% ε, του συνολικού παθητικού. Από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας σε επιμέρους εφημερίδες για το σκεπτικό πριν από το BRD, στην κρίση 2008-2011 μόνο σε μία περίπτωση αυτό το ποσό του 8% θα είχε πληγεί. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος ε, του κανονισμού και της οδηγίας αφορούν σαφώς στήριξη που δεν προέρχεται από τον δημόσιο τομέα, από το κράτος. Όπως ε, είπατε κι εσείς, αν τώρα πέραν από το bail-in του 8% του παθητικού, αν πέρα από το 5% του Ταμείου Εξυγίανσης, αν αυτά δηλαδή δεν επαρκούν, πρέπει βεβαίως να ε, βρούμε έναν μηχανισμό backstop, έναν ανασταλτικό μηχανισμό, ε, από το Ταμείο Εξυγείας πρέπει να προέρχεται. Υπάρχουν διατάξεις. Και από εκεί και πέρα, ενδεχομένως, προσωπική γνώμη βεβαίω αυτή, θα μπορούσαμε να αποτανθούμε στον μηχανισμό εποπτείας, στο ESM. Για να δούμε αν μπορούμε από εκεί να αποσπάσουμε κάποιους πόρους, μια στήριξη οικονομική, για να οργανώσουμε την εξυγίανση μιας τράπεζας. Ίσως υπάρχει τρόπος λοιπόν εδώ, αλλά όπως έχει υποθεί και σε διάφορα κείμενα, πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Είναι δύσκολο ζήτημα να βρούμε δηλαδή αυτή την λεπτή ισορροπία μεταξύ των επιμέρους οργανισμών, γιατί ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι το Ταμείο Εξυγίανσης αφορά μόνο τον τραπεζικό τομέα, ενώ ε, ο μηχανισμός εποπτείας αφορά την κρατική ενίσχυση και έχει απαραίτητα τον τραπεζικό κλάδο. Ευχαριστώ. Από πλευρά σοσιαλιστών, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε στην εισαγωγή σας Μιλήσατε για συντονισμό και συνεργασία. Αλλά είμαστε σε πενταγενές στάδιο μετά τον μηχανισμό ενιαίας εποπτείας. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς ακριβώς ε, θα διαμορφωθεί αυτή η συνεργασία και πώς μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα ε, κατά την ε, κατάρτιση του μηχανισμού εξυγείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα απαντήσω στα γαλλικά. Πράγματι, αυτό το ζήτημα της ε, συνεργασίας είναι κρίσιμη σημασία. αν θέλουμε να είναι επιτυχής αυτός ο μηχανισμός των δύο πυλώνων. Είναι σαφές ότι ο ενιαίος μηχανισμός παρακολούθησης εποπτείας θα έχει πραγματικά πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην πρόληψη των τραπεζικών κινδύνων. Και το βλέπουμε και στα κείμενα που υιοθετήθηκαν, στην οδηγία για την εξυγίανση. Και εκεί υπάρχει αυτό το ζήτημα της πρώιμης παρέμβασης που έχουν στη διάθεσή τους ε, οι αρχές εποπτείας. Και, ε, και στην Τραπεζική Ένωση έχουμε και το Συμβούλιο Εποπτείας. Τώρα, τι ακριβώς ε, θα κάνει το Συμβούλιο Εποπτείας. Ή μάλλον το, το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία ευθύς εξ από την ε, θέσπιση του ενιαίου ε, Συμβουλίου Εξυγίανσης και μετά. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί και να διαμορφωθεί απευθείας μια ομάδα εργασίας. Και νομίζω ότι και στις ε, προκαταρκτικές εργασίες του ε, προσωρινού Προέδρου ε, του Συμβουλίου αυτό ήταν μια προτεραιότητα. Μιλούμε λοιπόν για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο συμβουλίων δεν γίνεται να παρεμβούμε χωρίς να έχουμε δεδομένα, είναι λογικό. Και πρέπει να έχουμε δεδομένα και για την εξυγίανση και για την εποπτεία. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αξιοποιούμε αυτά τα δεδομένα και για τους δύο σκοπούς. Και μετά ο ίδιος ο μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων είναι το πρώτο βήμα μέχρι να περάσουμε στην εξυγίανση, που μετά γίνεται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οποίο είναι και πρακτικά, αλλά και πολύ πολιτικά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα εξετάσουμε εκ των προτέρων και μέσω μια ομάδα εργασία που θα πρέπει να ξεκινήσει εργασία τη ευθύ εξ αρχή. Ευχαριστώ, κύριο Σόρτσοκ από την ECR. Σα ευχαριστώ. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω να σα θέσω. Τι πιστεύετε για τις νέες προτάσεις σε ό,τι αφορά την δυνατότητα απορρόφησης των απολειών. Τι γίνεται με το υφιστάμενο σύστημα μεταρρύθμισης και πτώχευσης. Ε, sorry, I'm not sure to... Ε, Συγχωρέστε με. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτησή σας απόλυτα. Μιλάτε για τη χαμηλή απορροφητικότητα. Συγγνώμη, είχα κάποιο πρόβλημα κατανόησης. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχει το θέμα του να ξεκινήσουμε για τις ελάχιστες απαιτήσει για τις ε, ευθύνες αυτές. Για τα στοιχεία παθητικού. σε περίπτωση που χρειάζεται οργάνωση ε, bail-in. το, αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την σχηματισμό ενός πιο ανθεκτικού τραπεζικού κλάδου. Εκτιμάται ότι οι σημαντικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξέρουν ότι βασίζονται τα MRAIL στο σύνολο των μαθητικών στοιχείων. Ενώ σε διεθνέ επίπεδο η ιδέα ήταν να σχηματιστεί ένα σύστημα βασιζόμενο σε κριτήρια σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο χρέος. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά, γιατί θεωρείται ότι θα ήταν πιο κατανοητό σε διεθνές επίπεδο από τους ε, επενδυτές και από τις αγορές να υπάρχουν αυτά τα υφιστάμενα στοιχεία αντί για μία προσέγγιση η οποία ναι είναι θεωρητικά δυνατή αλλά πιο δύσκολα εφαρμόσιμη από το να αναγνωρίσουμε το δευτερεύον αυτό, το εφιστάμενο αυτό χρέος. τα Emrail, θα ξεκινήσουμε να τα υπολογίζουμε σε ό,τι αφορά τα ποσά που χρειάζονται οι τράπεζες δηλαδή του χρόνου και θα υπάρξει μια διεθνής πρόταση η οποία θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2016. Το ερώτημα λοιπόν για το Συμβούλιο και για εσάς είναι αν θα αναθεωρηθεί η οδηγία για να αντισταθμιστεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτός ο όρος για την απορροφητικότητα. Μέχρι το 2016 λοιπόν που θα οριστικοποιηθεί η πρόταση θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι χρειάζεται να το εφαρμόσουμε αυτό για κάθε τράπεζα σε ό,τι αφορά το MRAIL στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές ε, οι προδιαγραφές στις πιο συστημικά μεγάλες τράπεζες. Αυτά λοιπόν είναι κάποια ερωτήματα. Και δεν είναι τόσο απλό να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο όρων. Δεν είναι αδύνατον αυτό, αλλά εμπεριέχει την ανάλυση πολλών τεχνικών όρων. για να υπάρχει ένας πιο ανθεκτικός τραπεζικός κλάδος σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τράπεζες. Σας ευχαριστώ κύριος Γκίγκολτ. Ο προτινόμενος ε, τομέας ε, της ευθύνης και δεδομένου τα, των χαμηλών επιτοκίων που σημαίνει ότι παρά το γεγονός το οι τράπεζες ε, πληρώνουν ε, για το ε, ελάχιστο ή και για το μέγιστο χρέος, πώς μπορούμε να δεσμευτούμε οι τράπεζες να μπορούν πράγματι να εξηγιανθούν ώστε το πλεονέκτημα να μην υπάρχει για τις τράπεζες που είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν, για να πτωχεύσουν ε, επειδή αυτό στρεβλώνει την κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γίνει προγραμματισμός ώστε να αλλάξει η δομή και το μοντέλο το τραπεζικό, ώστε αυτή η γενής ε, ε, επιδότηση να μην είναι μία επιλογή. Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος, παρακαλώ πολύ. Απάντηση. Ε, σε γενικέ γραμμές πάντοτε θέλω να είμαι όσο το δυνατόν ε, πιο συγκεκριμένος. Αναφερθήκατε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Συμμετέχω σε διεθνή φόρα για τις συζητήσει αυτές ε, και είναι πραγματικά πάρα πολύ σαφές ότι οι συνθήκε της αγορέ σήμερα δεν μας δίνουν τη σωστή εικόνα του τιμήματος για τις τράπεζες ε, όταν ε, είναι πιο ανθεκτικές. Αυτό μπορεί να αφορά, να, είναι λόγω των ε, χαμηλών επιτοκίων. Βέβαια, το τίμημα δεν το πληρώνουν οι τράπεζες. Όταν εκδίδουν ομόλογα ή διάφορες άλλες υποχρεώσεις, με βραχυπρόθεσμη εγγύηση, 5-10 ε, χρόνια δηλαδή. Δεν ξέρουμε σε 5-10 χρόνια πώς θα είναι τα επιτόκια τα τραπεζικά. Οπότε και εδώ υπάρχει αυτό το οποίο εμείς ε, λέμε ε, προκυκλικότητα. Ένας κίνδυνος υποκατάστασης σε δύσκολες εποχές των υποχρεώσεων βάσει αυτής της δομής. Θέσατε το θέμα της ε, διάρθρωσης των, τραπεζών. υπάρχουν κάποιες μεγάλες τράπεζες ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ε, χώρες αυτές ε, υπάρχουν δύο διαστρωματώσεις, υπάρχουν εταιρείε καρτοφυλακίων, υπάρχουν οι τράπεζες και λόγω αυτής της διτής διάρθρωσης θα ήταν ευκολότερο να εκδίδει κανείς ομόλογα της εταιρείας χαρτοφυλακίου, ώστε να υπάρχουν ομόλογα εντός της τράπεζας ε, για να μπορούν να να γίνεται διάσωση με ίδια μέσα μέσω αυτών των ομολόγων. Αλλά αυτό ε, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά στοιχεία παθητικού, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ε, η δομή αυτή τύπου holding είναι η μοναδική δομή για να μπορούμε να έχουμε διεθνώς δραστήριες τράπεζες. Τώρα τι σημαίνει αυτό ως προς την δυνατότητα ε, εξυγίανσης. Αυτό βέβαια είναι το επίκεντρο της εξυγίανσης αυτής καθεαυτής. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα εξυγίανσης που να είναι αξιόπιστο αν δεν είναι εφαρμόσιμο. Οπότε το θέμα αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, την αντίκτυπο στις τράπεζες ε, μιας πιθανής εξυγίανσης. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα, πολλά υπέρ, πολλά κατά. Αλλά μόνο θέμα, ε, μόνο από την άποψη της, χρήσης του, της δυνατότητας χρήσης της διάσωσης με ίδια μέσα, του bail-in δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε το γεγονός ότι μία τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει μαζί με τα ε, διάφορα, με τις διάφορες, τα διάφορα υποκαταστήματά της. Αν συμπεράνουμε σε μερικές περιπτώσεις ότι θα πρέπει να αλλάξει η δομή, θα είχαμε τη δυνατότητα, θα είχαμε την εξουσία να το κάνουμε και είναι ακόμη μία φορά σαφές ότι η αξιολόγηση οι διάφορες απαιτήσει ε, προκειμένου να εξηγενθεί μια τράπεζα θα έπρεπε να, συζητηθεί, να και με τους υπεύθυνου εποπτείας. Ειδικότερα όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή ανησυχία για τις τράπεζες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Η Ντανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στα επιχειρηματικά μοντέλα, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε δει διαφοροποίηση των μοντέλων αυτών μεταξύ των τραπεζών και το επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι ουδέτερο θέμα από απόψεως εποπτείας αλλά και από απόψεως ε, εξυγίανσης. Όταν ε, κοιτάξει κανείς προς τα, προς τα πίσω τα τελευταία χρόνια, επειδή ήταν μια περίοδος κρίσης ε, και υπήρχε θέμα ανθεκτικότητας των τραπεζών έχετε εσείς ε, προτεραιότητα, ως προτεραιότητα το ένα ή το άλλο επιχειρηματικό μοντέλο, αν δει κανεί για παράδειγμα τις προκλήσεις που υπάρχουν σε σχέση με την εποπτεία και την εξυγίανση και το ερώτημά μου, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα εξυγίανση ε, τα οποία θα επεξεργάζεστε για πολύ καιρό και τα οποία ε, πρέπει να είναι στέρεα και χρειάζονται και πάρα πολλές επενδύσεις ε, εκατέρωθεν. Πιστεύετε ότι αυτά τα προγράμματα εξυγίανση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιο μελλοντοστραφέ εργαλείο στον τομέα τη Τραπεζικής Ένωση. ή μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι ένα εργαλείο ad hoc, το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια δεδομένη χρονική στιγμή σε περίπτωση που υπάρχει το χειρότερο δυνατό σενάριο. Τι διαρθρωτικά ζητήματα εκτός από το επιχειρηματικό μοντέλο ε, θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε με ένα στέρεο πρόγραμμα εξυγίανσης ή θεωρείτε ότι δεν είναι καθόλου αυτή η λύση που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των διαρθρωτικών ζητημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχα συνηθίσει να είμαι επόπτης για πάνω από 15 χρόνια. Δεν θα πω λοιπόν ότι η εξυγίανση είναι η λύση που θα, για όλα μας τα προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο, ανά τον κόσμο. Αυτό είναι σαφές, αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτή η διαδικασία εξυγίανσης, που είναι κάτι που μας απασχολεί σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και σε επίπεδο Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, θα μας παράσχει λοιπόν μια πραγματική αλλαγή στον τραπεζικό κλάδο για, τους, για τα πιο σημαντικά θεσμικά όργανα. Μπορείτε να δείτε ότι σε κάποιες ε, χώρες μεγάλες τράπεζες πουλούν περιουσιακά του στοιχεία, πουλούν θηγατρικές και εδώ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακατατάσσουν, αναδιαμορφώνουν τις ε, δραστηριότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι η εξυγένση δεν είναι το τέλος. Ο σχεδιασμός εξυγένσης θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον και σημαντικό μέσο για να ενισχύσουμε, να έχουμε πιο ανθεκτικές ε, τράπεζες. Θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε τις κρίσιμες σημασίες λειτουργίας. λειτουργίες. Από πλευρά εξυγίανση, λοιπόν, το σημαντικό είναι τι εξουσία μπορεί να έχει η αρχή εξυγίανση να αποδεσμεύσει κάποια στοιχεία μια τράπεζας και να τα θέσει σε μια άλλη και ούτω καθεξή. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πραγματική ανάγκη οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων εντός των ε, επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών. Προς το παρόν Κάποιες τράπεζες έχουν πολύ ε, διαφορετική δομή. Εφόσον ε, μιλάμε και για οικονομίες ε, κλίμακας. Από πλευρά εξυγίανση, λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να είναι πιο σαφή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ακόμα και να ζητήσουμε αλλαγές τη δομή της λειτουργίας ακόμα και στο εσωτερικό μίας ε, τράπεζας και των επιμέρους επιχειρηματικών γραμμών. Αν υπάρχει κάποιο καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο. Δεν είμαι σίγουρος ότι η αρχή εξυγίανσης ε, έχει αυτό το ρόλο. Να πούμε δηλαδή ποια είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν θέλουμε να κρίνουμε δεχόμαστε την πραγματικότητα όσο έχει αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο αυτό το Ίδρυμα ε, είναι δυνατόν να εξηγενθεί ή όχι από πλευράς προστασίας ε, καταθέσεων, μη αξιοποίησης δημοσίων πόρων, χρηματοοικονομικής σταθερότητας και διατήρησης αυτών των περίφημων κρίσιμων λειτουργιών είναι ζήτημα εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο και στην ικανότητά του να χρηματοδοτεί την οικονομία. Και όχι τόσο ε, τη διατήρηση ενός ε, επιχειρηματικού ε, μοντέλου επάπειρων. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πράγματι λοιπόν τα σχέδια εξεγείανσης θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο αλλαγής του τραπεζικού κλάδου Νομίζω ότι το σχέδιο εξυγίανσης θα πρέπει να καταρτίζεται σε βάση ad hoc, γιατί και πάλι εμείς εδώ δεν είμαστε εδώ για να σας δώσουμε μία γενική λύση για όλες τις τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κομμένο και ραμμένο το κάθε πρόγραμμα στην κάθε τράπεζα, αλλά είναι κάποιες διαφορετικές αλλαγές που τις χρειάζονται περίπου όλες οι τράπεζες. Ωραία. Ε, ζητώ από όλους τους ομιλητές να μείνουν στα πέντε λεπτά. Ο κύριο Μόνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Δύο ερωτήματα. Αρχικά, το τραπεζικό παράδοξο, όπω το αποκαλώ. Λέμε ότι τα stress test για τους συστημικούς κινδύνους ε, είχαν οικονομητικά αποτελέσματα. Αυτό Μα εξήγησε ο κύριο Δράγκη η κυρία Νούη στις, στα τέλη Οκτωβρίου, αρχέ Νοεμβρίου. Και από την άλλη θεσπίζουμε μια τραπεζική ένωση με τραπεζική εποπτεία συν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση και το συμβουλίο τη. Εσεί θεωρείτε ότι η τραπεζική εποπτεία αρκούσε Μήπως θεωρείτε λοιπόν ότι αρκούσε, γιατί ήδη υπήρχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε stress Δεύτερον, α πούμε ότι υπάρχει ένα υποθετικό σενάριο. Μία μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα, τη Ευρωζώνη τουλάχιστον, υπό την εποπτεία τη ΕΚΤ, πτωχεύει. Α υποθέσουμε το χειρότερο σενάριο. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε, για παράδειγμα, στην Γαλλία, τα τρία πρώτα βήματα που θα κάνατε για ένα σχέδιο εξυγίανση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα. το βάθος ε, της κρίσης την οποία περίλθαμε από το 2008 και μετά ε, δεν εκλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που έγινε πολύ πιο βαθιά αντιληπτό σε κάποιες χώρες που είδαν το τραπεζικό του σύστημα πραγματικά να ισοπεδώνεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το βάθος της κρίσης. Κάτι που δεν ισχύει σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία που κατάφεραν ε, να θεωρήσουν τουλάχιστον ότι το, σύστημα, το τραπεζικό του σύστημα ήταν πιο ανθεκτικό. πέραν λοιπόν μια τέτοια ε, κρίση, τέτοιου μεγέθους και τέτοιου βάθους στην Ευρώπη, που ακόμα και σήμερα μας επηρεάζει, εμάς τους Ευρωπαίου πολίτε. Βέβαια και με την ε, δημόσια στήριξη που έπρεπε να παρασχεθεί, Έπρεπε λοιπόν και να δώσουμε μια σειρά απαντήσεων. Χρειαζόταν εμπιστοσύνη. Είναι θεμελιώδε αυτό το στοιχείο. Αυτή η εμπιστοσύνη λοιπόν βασίζεται, όπως είπα και εισαγωγικά, στην εξέλιξη της ε, νομοθετικής εξουσίας και των θεσμικών οργάνων. Σε αυτό το επίπεδο, εσεί ω ε, θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή, κάνατε εξαιρετική πρόοδο σημειώσατε για να ε, επιφέρετε σημαντικές βελτιώσεις αυτούς τους δύο άξονες. Και στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες λοιπόν και από πλευράς μέσων ε, εποπτεία και εξυγίανση ταυτόχρονα. Τα stress test ήταν θετικά και όλοι είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Ε, αυτό αποδεικνύει μάλιστα ότι πολλά έχουν ήδη γίνει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τα ζητήματα εποπτείας και επιπλέον εξυγίανση. για να ξεκινήσουμε από μια εύρωστη βάση κατόπιν αυτών των stress test, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. Αν μπορούμε να μείνουμε στην εποπτεία. Απολύτως όχι. Νομίζω ότι η εξυγίανση μας δίνει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, με πολύ σημαντικές εξουσίες και μέσα, ακριβώς για να εγγυηθούμε τις ε, καταθέσεις, να διασφαλίσουμε το σύστημα και έτσι το οπλοστάσιο ε, που έχει τεθεί στη διάθεση του ε, Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι πολύ δυνατό για να διασφαλίσει ακριβώς το μέλλον του τραπεζικού κλάδου προ όφελο τη ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, όπω είπατε, αν πτώχευε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα, τι θα κάναμε. Πρώτα, θα έπρεπε να δούμε εάν αυτή η πτώχευση ε, απαιτεί να μπούμε σε στάδιο εξυγίανσης. Αν δηλαδή πρέπει να πούμε ότι θα τις ε, σώσουμε όλες τις τράπεζες. Όχι. Και οι επιχειρήσει, ε, συγγνώμη, και οι τράπεζε επιχειρήσει είναι όπως οι υπόλοιπε. Εντάξει, έχουν διαφορετική λειτουργία, αλλά το πρώτο βήμα θα, είναι, θα ήταν να επαληθεύσουμε ότι είναι απαραίτητο να μπούμε σε φάση εξυγίανσης για να διασφαλίσουμε τις κρίσιμες λειτουργίες και την οικονομική σταθερότητα και το καθεξής. Από τα πρώτα βήματα λοιπόν θα ήταν να εμπνευστούμε από το σχέδιο εξυγίανσης που θα είχαμε στη διάθεσή μα, αλλά πρέπει να δούμε αν ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη κρίση την οποία αντιμετωπίζει αυτή η τράπεζα. Ίσως θα πρέπει να το προσαρμόσουμε. Μετά υπάρχει και μια αλλαγή διοίκηση, σίγουρα. Και μετά η διατήρηση των κρίσιμων λειτουργιών με μια ε, συμπληρωματική τράπεζα ε, με την διάσωση με ιδίους πόρους, bail-in. Έτσι, για να σας τα πω σχηματικά, λαμβάνουν δράση τα θεσμικά όργανα, μετά μοιράζουμε, βλέπουμε τι ακριβώς είναι απαραίτητο και τι μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρο και διάσωση με ίδια μέσα. Είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε μεταξύ άλλων. Επερώτηση. Διακόπτει ο πρόεδρος. Για 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε... Λυπάμαι, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε και άλλους υποψηφίους και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Σίμων, τελευταίος ομιλητής. Δύο ερωτήσει έχω να σας θέσω. Δύο ερωτήσει, λοιπόν. Καταρχάς, σε σχέση με τα εθνικά συστήματα και με την Τράπεζα ενισχύσεων. Έχουμε την ε, δυνατότητα μέχρι 50% να χρησιμοποιήσουμε εθνικά μέσα για τους πόρους. Στην ε, φάση λοιπόν οικοδόμησης του συστήματος του SRM ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αν είναι ακόμα μικρό λοιπόν το Ταμείο Εξυγίανσης, υπάρχει μεγάλος πειρασμός να βγει το 50% από τους εθνικούς πόρους. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρχει συντονισμός με τα εθνικά, με τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες, προκειμένου να διατηρηθεί και το εθνικό σύστημα αλλά και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας, προκειμένου να υπάρχει και σταθερότητα. Δεύτερο ερώτημα για τις τράπεζες. Υπάρχουν πολλές τράπεζες που έχουν εθνικές εγγύησεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα πτώχευσης γιατί μπορεί να είναι πιο χρήσιμη, πιο ωφέλιμη η εξυγίανση των τραπεζών αυτών ή τμήματων των τραπεζών αυτών. Ποια είναι λοιπόν η σχέση των δημοσίων, των αθνικών αρχών και των δικών σας αρχών που θα μπορούσαν ενδεχομένω να παρέμβουν και να πούν ότι όχι, δεν θα γίνει εξυγίανση, δεν θα γίνει διάσωση με εθνικούς πόρους. Μπορείτε να φανταστείτε μια κατάσταση τέτοια. Η απάντηση. Σύντομη απάντηση, αν θέλετε, λέγει ο Οι σχέσεις με τα συστήματα εγγύησης ε, καταθέσεων. Σωστά λέτε ότι τα συστήματα αυτά είναι ένα βασικό στοιχείο για να δοθεί εμπιστοσύνη στους καταθέτες. Η οδηγία για το BRD για την ανάκαμψη και την εξυγένση, όπως την ερμηνεύω εγώ. Τι λέει, ότι μπορεί να υπάρχει παρένδυση για την αντισταθμίση, των ε, απώλειων, όχι για να επανακεφαλαίωση απαραίτητα, προστασία των καταθέσεων, λοιπόν, Το δεύτερο λοιπόν σύστημα εγγύησης καταθέσεων προβλέπει ένα ποσό. Σε εθνικό επίπεδο κάθε φορά, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία πρόσθετη προστασία των κατάθετων. Σε κάποιες χώρες, δεν να προσθέσω, υπάρχει δυνατότητα το σύστημα καταθέσεων εξάντε να παρεμβαίνει και όχι απαραίτητα τη στιγμή της εξυγίανσης. Τι διαδραματίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των τραπεζών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Έχετε δίκιο λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει η σωστή αλληλεπίδραση, η σωστή σχέση όπως ε, βλέπετε στην οδηγία, οι εκπρόσωποι των ηθήνων αρχών μπορεί να είναι μέλη του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Δηλαδή, η ομάδα συνεργασίας και η συνεργασία η ίδια ήδη κατοχυρώνεται στο κείμενο και όταν υπάρχει λοιπόν, όταν θα έχουμε στα χέρια μας τους κανόνες, θα μπορέσουμε να του διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυηθούμε τη συνεργασία. Για τη δεύτερη ερώτησή σα. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνε. Η εξυγίανση των τραπεζών. Ακόμα και όταν υποτίθεται ότι γίνεται για να αποφευχθεί η δημόσια στήριξη, δεν θα αλλάξει την κατάσταση πριν την κρίση. Το γεγονός λοιπόν ότι δόθηκε δημόσια στήριξη σε μία τράπεζη μετά από εξέταση φυσικά από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού όλα αυτά θα μπορέσουν να διατηρηθούν σε κάποιο βαθμό. Η ιδέα είναι να διατηρηθεί η κρίσιμη λειτουργία και τα στοιχεία που είναι κεντρικά για να υπάρχει ένα σύστημα τραπεζών που δεν θα έχει αντίκτυπο στις άλλες τράπεζες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το εμπόριο, είναι σημαντικό να μην υπάρχει αντίκτυπος υπερχείλησης αν θέλετε και επιρροής άλλων συναλλαγών σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι οι στόχοι της ε, οδηγίας. Να αντιτηρηθεί η σταθερότητα προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση περισσότερων δημοσίων πόρων και να μην υπάρχει αντίκτυπος ε, στους, στα άλλα ιδρύματα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ακρόαση. Και κλείνει λοιπόν το σημείο αυτό. Και περνάμε στον επόμενο υποψήφιο. Uh, Καλωσορίζουμε τον κύριο Αντώνιο Καρασκόζα, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής ε, της ε, ε Ισπανικής Αρχής ε, για τη σωστή αναδιάρθρωση των τραπεζών. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας για την επίσημη αυτή ακρόαση. Συγχαρητήρια για ε, την ε, υποψηφιότητά σας. Ε, σας διόρισε υποψήφιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, Διευθυντή Προγραμματισμού Εξυγίανσης ε, του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ε, Έχουμε ήδη κάνει μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Καρασκόζα. Σας καλωσορίζουμε, χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Μεταδίδεται η συνεδρίασή μας και στο διαδίκτυο, ζωντανά. Σας δίνω το λόγο για εισαγωγικά σχόλια Πέντε λεπτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και ε, συγκεκριμένα ε, είναι τιμή μου η σημερινή ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της οδηγίας όπως επίσης και του κανονισμού για την τραπεζική εξυγίανση. Μεγάλη χαρά λοιπόν για μένα να βρίσκομαι εδώ. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου για πλήρες ε, μέλος ε, του ε, Συμβουλίου Εξυγίανσης. Πρόκειται για ένα συμβούλιο το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ενιαίου, συστήματος, του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης είναι ένα βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης. Ε, εγώ έχω άμεση εμπειρία ε, της ε, Τραπεζικής Ένωσης στην Ισπανία. Ήταν αδύνατον στη χώρα μου πριν από δύο χρόνια να γίνει η σύνδεση, η στρεβλή σύνδεση μεταξύ του ε, τραπεζικού ε, χρέους και του ε, κρατικού χρέους. Και αυτό είναι ένας βασικός σκοπός του, της Τραπεζικής Ένωσης, είναι να διατηρήσει την, τον τραπεζικό τομέα και την αποφυγή της σύνδεσης αυτών των δύο πραγμάτων που ανέφερα προηγουμένως ο βασικός στόχος του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης είναι η αποφυγή της ε, χρήσης ε, των ε, δημοσίων κεφαλαίων για τη διάσωση των τραπεζών. Μέχρι τώρα, σε όλες τις κρίσεις του τραπεζικού τομέα, δημόσιο χρήμα έχει χρησιμοποιηθεί εξού και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής. Έχουμε τώρα πλέον μία διαφορετική προσέγγιση που βασίζεται στο bail-in των ε, οικονομικών ε, μέσων, οπότε θα υπάρχει ανακεφαλαιοποίηση λεπτομερής, που θα ρυθμίζεται σε λεπτομερές επίπεδο και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε, ελπίζουμε, τις διασώσεις στον τραπεζικό τομέα. Ένας ακόμη στόχος του μηχανισμού αυτού είναι να αποφύγει την ε, οικονομική έλλειψη ε, σταθερότητας, ε, την έλλειψη οικονομικής σταθερότητας μετά που διαπιστώνεται κρίση σε μία τράπεζα. Και στη χώρα μου έχουμε εμπειρία ε, της τραπεζικής πίστοσης, της έλλειψης τραπεζικής πίστοσης ε, μετά ε, την σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση που υπήρξε στην Ισπανία. Είναι λοιπόν ε, εκτενής η εμπειρία μου στον ε, τομέα της εξυγίανσης. Έχουμε εξυγιάνει εννέα τράπεζες στην Ισπανία. Ε, το ενεργητικό τους είναι περίπου 65 με 70% του ισπανικού ΑΕΠ. Οπότε μιλάμε για, ένα για μια σημαντική χρηματοπιστωτική κρίση. Θα αξιοποιήσω όλη την εμπειρία μου για να προσπαθήσω να εφαρμόσω ορθά τον ε, κανονισμό, ε, όλους τους κανονισμούς, ε, τους συναφείς με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το bail-in είναι κάτι το οποίο υπάρχει επί χάρτου, υπάρχει στο νόμο, αλλά πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειές του. Πρέπει να δούμε τον τρόπο ε, εφαρμογής αυτού του νέου μοντέλου. Αυτού του νέου μοντέλου. Οπότε είναι ευπρόσδεκτη όλη η προσπάθεια των ευρωπαϊκών οργάνων για την λεπτομερέστερη διαμόρφωση του συστήματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ο κύριος Ζάλμπα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασκόσα για την εισήγησή σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και πάλι εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την πείρα σας. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό, Ήσασταν ένας από τους λίγους που είχατε κάποια πείρα στην εξυγίανση. Είστε ειδικό στην εξυγίανση λοιπόν. Βάσει αυτής της εμπειρίας λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε μάθει από όλη τη διαδικασία. Θα ήταν χρήσιμο αυτό για τις νέες ε, αρμοδιότητες που θα λάβατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση μεταξύ των γενικών διδαγμάτων που μπορούμε να αντλήσουμε από μια εμπειρία και των διδαγμάτων που συνδέονται συγκεκριμένα με τα μέσα εξυγίανσης. Σε ό,τι αφορά τα γενικά διδάγματα, πολλά έχω μάθει. Πρώτα απ' όλα, η σημασία της ε, της δυνατής ε, ανάλυσης της κατάστασης, μιας ε, τεκμηριωμένης βέβαια αντικειμενικής ανάλυσης ε, της κρίσης στο τραπεζικό σύστημα. Στη χώρα μας αυτό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ε, είχαμε μπερδέψει το πρόβλημα ρευστότητα με το ζήτημα της ε, φερεγγιότητας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η διάκριση των των δυνατών γιατί η δάλος το κόστος της επίλυσης του προβλήματος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Η ανάλυση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, Από την εμπειρία μου λοιπόν, μίλησα για την ε, σημασία της ανάλυσης ε, και αυτό, αυτό το stress test και πόσο σημαντικό είναι να γίνονται όλα αυτά ανεξάρτητα. Εμείς είμαστε υπέρ της εξαγωγής stress test και αναθεώρησης πέραν ε, της εποπτικής αρχής και γι' αυτό και έχουμε προσλάβει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να διεξάγουν ακριβώς αυτά τα stress test. Και έχουμε λάβει τέτοια εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και από την ΕΚΤ και από άλλους φορείς. Άλλο ε, δίδαγμα τώρα είναι η αναγκαιότητα εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών κατά τη διάρκεια των τραπεζικών κρίσεων. Στην Ισπανία είχαμε δύο εναλλακτικέ. Μία το 2011. Εκεί ζητήσαμε κεφάλαια από τις ίδιες τις τράπεζες και είχαμε θεωρήσει ότι αυτό θα αρκούσε ότι εκείνε δηλαδή θα μπορούσαν να εξηγειάνουν τους ισολογισμού τους. Όμως αυτό απεδείχθη λανθασμένη εκτίμηση και το 2012 τελικά δαγκαστήκαμε να τις αναγκάσουμε στην εξυγίανση για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το κίνδυνο. Να τις εξηγιάνουμε λοιπόν και να μην αφήσουμε τις τράπεζες να κάνουν την εξηγίανση μόνες τους. Και τέλος, ό,τι αφορά τη μακροοικονομική κατάσταση, είναι πολύ πιο εύκολο να επιλύσει κανείς ε, μια τραπεζική κρίση όταν η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται. Όπως στη Σουηδία, για παράδειγμα, αν δείτε τη δεκαετία του 90. Και αυτό ήταν μια παράδειγμα εύρυθμης λειτουργίας, καλής διαχείρισης της τραπεζική κλίση, όμως ε, εποφελήθηκαν και μια ε, γενική οικονομική ανάκαμψη. Σε ό,τι αφορά το, τη διάσωσε με ίδια μέσα, το bail-in, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και καλή εμπειρία των χρηματοκο... εμπορία των χρηματοοικονομικών μέσων. Γιατί οι επενδυτές αυτών των μέσων θα αναλάβουν τμήμα του βάρους της αναδιοργάνωσης και της εξυγίανσης. Αυτό συνέβη και στη χώρα μου. Είχαμε είχαμε πολλές δικαστικές διαφορές εξαιτία της κακής εμπορίας αυτών των προϊόντων. Και τέλος, ε, για τους φορείς αυτούς, αυτά τα ιδρύματα, είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση να μην είναι βιαστική. Πρέπει να αναλύει την κατάσταση, να εξετάζει εναλλακτικέ λύσεις και μετά να ενεργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην περίπτωσή μας είδαμε το σύνολο των ιδρυμάτων, αφαιρέσαμε τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, εξετάσαμε διάφορες στρατηγικές, όμως το καλύτερο είναι να μην βιάζεται κανείς, γιατί τότε μπορεί να οδηγηθεί σε υψηλότερο τελικό κόστος. Και τέλος, για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ε, μιας Κακή τράπεζα αν ε, όπως την αποκαλούν. Τώρα, κατά πόσο θα πρέπει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν σε μια, ε, προβλήματα, ε, σε μια τράπεζα που έχει προβλήματα. Πρέπει να τα αφαιρέσουμε και να μεταφέρουμε να τα μεταβιβάσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία σε μια επιχείρηση, σε μια τράπεζα που χειρίζεται ακριβώς ε, αυτά τα στοιχεία και αυτό ήταν μια καλή επιλογή. Ευχαριστώ κύριο Μπαγιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καρασκόσα που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα. Όπως είπατε και εσείς, είναι σημαντικό οι τράπεζες να ε, περνούν σε διάσωση με ίδια μέσα και όχι σε bailout, αλλά είδαμε και με τα stress test ότι κάποιες τράπεζες ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εσείς ε, τι μέτρα θα μπορούσατε να πάρετε για να ε, θεσπιστεί γρήγορα το Συμβούλιο Εξυγίανσης και να μην βρεθούμε και πάλι στην κατάσταση ανάγκης χρηματοδότησης τραπεζών. Μετά και πάλι για το stress test. Μιλάμε για σταδιακή ανακεφαλαιοποίηση. Τι συμβαίνει λοιπόν εάν ε, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να υιοθετηθούν στους επόμενους μήνες. Ποιο βαθμό αντίδραση θα μπορούσε να καταστεί επιχειρησιακό. Και εσεί τι θα κάνατε για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ταχύτατα προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε το στομότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία της οδηγίας και του κανονισμού. Ακόμα και χωρίς τον καινούργιο κανονισμό, στην χώρα μου για παράδειγμα, εφαρμόσαμε το σύστημα του bail της ε, διάσωσης μέσα. Στην Ολλανδία επίσης οι αρχές έχουν εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές Έχουμε λοιπόν την εμπειρία να το κάνουμε αυτό. Άμεσα μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για να ξεπεράσουμε μια τραπεζική κρίση πριν την πλήρη εφαρμογή. Την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας και του κανονισμού. Για το μέλλον δε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ του σχεδίου εξυγίανσης εξάντε και της σχετικής αξιολόγησης. Θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση του πώς μπορούμε να κάνουμε εξυγίανση τραπεζών μικρών και μεγάλων. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς δημόσιους πόρους. Αυτό θα πρέπει να είναι τελευταίος, να είναι η τελευταία διέξοδος. Στη χώρα μου έχουμε κάνει κάποια τέτοια δουλειά και εφαρμόζοντας τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφύγαμε όλο το ποσό που είχε μπει στο τραπεζικό σύστημα το 2012 50 εκατομμύρια ευρώ και είχαμε μεγάλα ιδρύματα από συμπάνκια, αλλά και μικρά ιδρύματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει όλα αυτά τα ιδρύματα να εφαρμόσουν την οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά το σχέδιο διάσωσης εξάντε να είμαστε επίσης ε, φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες απαιτήσει για επιλέξιμες υποχρεώσεις, τα MREL, και έτσι είμαι βέβαιος ότι θα αποφύγουμε να χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα στο μέλλον για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Σοζόκα από τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Ευχαριστώ πολύ. Μία συγκεκριμένη ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και για την σωστή εξυγίανση και σε ό,τι αφορά τα δευτερεύοντα χρέη. Πώς θέλετε να συνεργαστείτε με τις εθνικές αρχές πώς σκοπεύετε να τηρήσετε όλες τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη θέση σας. Βράχει πρόθεσμα. Νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι η σύσταση του θεσμικού οργάνου με όλες τις εξουσίες που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί μια τραπεζική κρίση. Μακροπρόθεσμα τώρα. Πιστεύω ότι η πρόκληση έγκυται στο πώς θα καταστεί αξιόπιστο το εργαλείο του Μπέιλιν. Προκειμένου να μην υπάρχει συμμετοχή δημόσιου χρήματος. Διάβασα χθε την έκθεση της ε, Moody's του Οργανισμού Αξιολόγησης Επιστρεπτικής Ικανότητας που αναφέρει ότι δεν εμπιστεύεται την διαδικασία του bail-in, της διάσωσης με ίδια μέσα. Ο κόσμος προτιμάει το bail-out με τα χρήματα του φορολογούμενου. Προφανώς, γιατί δεν χρειάζεται να βάλει ειδικού του πόρους. Αλλά αν στο μέλλον θέλουμε να αποφύγουμε χρήση δημοσίων πόρων, θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι στο σχέδιο εξυγίασης εξάντε. Γιατί στην παρούσα φάση η αντιμετώπιση του προβλήματος μιας τράπεζας είναι πολύ πιο δύσκολη. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σκληρά για τα σχέδια εξυγένσης εξάντε και θα πρέπει να πούμε και να δείξουμε στις αγορές ότι είναι και εφικτό αλλά και σωστό το νέο εργαλείο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του νέου μοντέλου, θεωρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η από την Άλντε. Καλημέρα σας κύριε Καρασκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ θα ήθελα ένα πράγμα να σας ρωτήσω. Μιλήσατε ορθά ε, για ε, το κανονισμό του μηχανισμού. Ε, εμείς συμμετείχαμε, οπότε τις γνωρίζουμε. Είπατε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αξιοπιστία. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για το θέμα ευρωζώνη και εκτός ευρωζώνης. Τι θα γίνει στην περίπτωση εποπτείας ε, για τις χώρες της Ευρωζώνης, πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε το μην κατακαιρματισμό της αγοράς. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε και ξέχασα την τελευταία ερώτηση να απαντήσω τη συνεργασία με τις εθνικές, εποπτικές, συγγνώμη, με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης χρειάζεται ένα ισχυρό συμβούλιο εξυγίανσης και χρειάζεται και σαφής συντονισμός ε, με ε, το, την Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα όπως επίσης και με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, γιατί τουλάχιστον πρόθεσμα εμείς βασιζόμαστε στις εθνικές αρχές εξυγίανσης με άλλους τώρα ευρωπαϊκούς παίκτες. Η, η συνεργασία είναι βέβαια μεγάλη σημασίας και με την Ευρωπαϊκή Αρχή, Τραπεζική Αρχή, την EBA, για το θέμα των απαιτήσεων για επιλέξιμες υποχρεώσεις ε, είναι ε, σημαντική η συνεισφορά τους. Έχουν ε, δημοσιεύσει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο προσπαθεί να ε, προτείνει τρόπους εφαρμογής του ΕΝΡΕΛ. E Για τις χώρες βέβαια εκτός ε, Ευρωζώνης, ο συντονισμός είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η συνεργασία. Στην περίπτωση διασυνοριακών ε, οργανισμών. Έχουμε πολύ σημαντικούς διασυνοριακούς οργανισμούς. Για την ώρα υπάρχει ένα, υπάρχουν εθνικά πλαίσια εξυγίανσης, οπότε χάρη στη νέα οδηγία και στο νέο κανονισμό έχουμε ένα στέρεο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το Συμβούλιο Εξυγίανσης, και με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης έχουμε το ρόλο των σωμάτων εξυγίανσης ε, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, της EBA, που προσπαθεί να μεσολαβήσει σε περίπτωση ε, προβλημάτων εξυγίανσης. Έχουμε λοιπόν ένα καλό πλαίσιο, κατά την άποψή μου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, της εξυγίανσης των τραπεζών στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Σβέν Κίγκολ. Μας απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι το τίμημα για τα μικρότερα για τα χαμηλότερα και τα υψηλότερα ομόλογα είναι ε, ιστορικά ε, χαμηλό. Ε, υπάρχει πολλής λόγος που γίνεται, πάρα πολύ νομοθεσία. Ε, έχουμε ε, κάνει ε, υπολογισμού και τα έχουμε λάβει όλα υπόψη. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν προγράμματα εξυγίανση που να εξασφαλίζουν ότι υπάρχει αξιοπιστία του bail-in. Μήπως μπορείτε να μα πείτε λοιπόν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα ποιε αλλαγέ στα επιχειρηματικά μοντέλα και στη διάρθρωση των τραπεζών θα προωθήσετε προκειμένου το bail-in να είναι αξιόπιστο και για τις αγορές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πράγματι αξιόπιστο το, το γεγονός ότι έχουν χίλιες υποκατα, χίλια, υποκαταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο οι τράπεζες και αυτό δεν καθιστά ευκολότερο το bail-in και την εφαρμογή πραγματικών εργαλείων εξυγίανσης. Παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος. Πώς μπορούν να αλλάξουν οι τράπεζες, πώς πρέπει να αλλάξουν ώστε να είναι αξιόπιστη η διαδικασία του bail-in. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διαρθωτικά μοντέλα. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως γνωρίζετε. Το ενιαίο σημείο εισόδου και το πολλαπλό σημείο εισόδου. Single και multiple point of entry. Στην περίπτωση της Ισπανίας, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε το πολλαπλό σημείο εισόδου. Στη Σανταντέρ, για παράδειγμα, Έχουμε 10 αποκαταστήματα στο εξωτερικό. Και έτσι θα έχουμε και 10 φορείς εξυγίανσης. 10 διαφορετικούς φορείς λοιπόν που θα εφαρμόσουν τη διάσωση με ίδια μέσα. Για εμάς λοιπόν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη αυτή η προσέγγιση. Αλλά έχουμε και την πλειονότητα των συστημικών τραπεζών που ακολουθούν την προσέγγιση του ενιαίου σημείου εισόδου. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μόνο μία αρχή εξυγίανσης. Την μητρική εταιρεία. Και εκεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη διάσωση με ίδια μέσα σε αυτό τον ενιαίο φορέα του ομίλου. Από τη δική μου εμπειρία λοιπόν, το πολλαπλό σημείο εισόδου μπορεί να είναι η κατάλληλη εναλλακτική λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, να μην έχουμε εκατοντάδες ε, υποκαταστήματα ανά τον κόσμο και έτσι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με αξιόπιστο τρόπο το bail-in. Άλλες διαθετικές αλλαγές. Περισσότερο τώρα στο πεδίο των προληπτικών μέτρων. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή για τον ε, διαχωρισμό των επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών. Υπάρχει τέτοια συζήτηση και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ευρωπαϊκό Βασίλειο. Αλλά μάλλον όλα αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια αποφυγής τέτοιας χρηματοπιστικής κρίσης στο μέλλον. Επομένω, το ερώτημά σας θα έλεγα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο, στη συζήτηση της επιλογής μεταξύ πολλαπλού και ενιαίου σημείου εισόδου. Ευχαριστώ. Η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω για το εξής. Οι εθνικοί κανόνες και οι εθνικοί νόμοι αφαιρεγγιότητας και σχετικές διαδικασία δεν είναι συντονισμένοι και εναρμονισμένοι. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει το έργο σας η Εθνική Νόμη για την αφαιρεγγιότητα και οι εθνικές δραστηριότητες και διαδικασίες. Αυτό θα επηρεάσει το έργο σας στο ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης με το πλαίσιο εξυγίανσης προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την εφαρμογή των κανονικών κανόνων και διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. Αν λοιπόν με επιτυχία εφαρμόσουμε τα εργαλεία εξυγίανσης, φυσικά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα σε κάποιες ε, χώρες όταν θα χρειαστεί να εφαρμόσουν την εξυγίανση. Αλλά από πλευράς γενικής, ο μηχανισμός εξυγίανσης και ο κανονισμός για την εξυγίανση προσπαθεί ακριβώς να αποφύγει την εφαρμογή των κανονικών διαδικασιών και νομοθεσιών αφαιρεγγιότητας. Μπορεί να εμφανιστούν κάποια ίσονο σημασία προβλήματα, αλλά αν με επιτυχία εφαρμόσουμε την προσέγγιση της εξυγίανσης, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο τελευταίος ομιλητής τώρα. Στα γερμανικά θα σας θέσω το ερώτημα. Μία ερώτηση, την οποία προηγουμένως θέσα και στους προηγούμενους υποψήφιους. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας απάντηση. Σχέση των συστημάτων ασφάλισης με τους μηχανισμούς εξυγίανσης. Έχουμε λοιπόν το σύστημα με τους ε, πιστωτές, έχουμε και το στέλος ε, το ταμείο, αλλά υπάρχει ενδιάμεσα μία δυνατότητα bail-in μέχρι 50% των χρημάτων. Και αυτό καλώς έχει. Αλλά στη φάση όπου το Ταμείο Εξυγίανσης οικοδομείται και στο εθνικό σύστημα υπάρχουν πιο πολλά χρήματα, μπορεί να μην φτάσει το bail-in με ίδια μέσα δηλαδή και στο ταμείο δηλαδή να μην υπάρχουν αρκετά μέσα. Και έτσι λοιπόν να υπάρχει κίνδυνος παρέμβασης των εθνικών ε, εργαλείων. Αλλά αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε κατάρρευση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Έχουμε το μηχανισμό εξυγίανσης αφενός με, τα, την ευρωπαϊκή ιδιότητα, από την άλλη έχουμε τα εθνικά συστήματα και κατά τρίτον έχουμε την υποπτική αρχή στην Φραγκφούρτη, η οποία ενδεχομένω να έχει πάλι άλλα μέτρα και σταθμά. Ακούσατε ποια ήταν η απάντηση του προηγούμενου υποψηφίου. Όντω υπάρχει εκπρόσωπό σα ε, που συμμετέχει, αλλά σε περίπτωση διαφωνίας. Ποιος θα λάβει τελικά την απόφαση. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα διαμορφωθεί μια τέτοια κατάσταση κάποια στιγμή. Η απάντηση. Νομίζω ότι αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα θετικών εγγυήσεων θα έχουμε ένα πρόβλημα. πρώτα λοιπόν από ό,τι ξέρετε θα πρέπει να βασιστούμε στο bail στην διάσωση με ίδια μέσα για το κεφάλαιο, για τα παλαιά χρέη. Για την Ισπανία για παράδειγμα. Αυτό θα μπορούσε να σήμαινε επίλυση των προβλημάτων. Έχουμε συστημική κρίση στο χρηματοπιστωτικό μας ε, σύστημα. Στις καταθέσεις θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μη καλυπτόμενες καταθέσεις. Να περάσουμε στη συνέχεια στις καλυπτόμενες καταθέσεις. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία πολύ σύνθετη και παραπάνω από συστημική τραπεζική χρήση, αλλά όπως είπατε, το σύστημα εγγύησεων καταθέσεων μπορεί να καλύψει μέχρι και 50% του στόχου χρηματοδότησης. Συνολικά λοιπόν πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης τραπεζικής κρίσης. στην Ευρώπη. αν χρειαστεί να εφαρμοστούν οι υποθνικοί τρόποι εφαρμογής ε, της εξυγίανσης, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Του Υπουργείου Οικονομικού, τα χρήματα του ESM με διάφορες δυνατότητες, έχουμε θέματα κεφαλαιοποίησης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σταθερό το πλαίσιο που υπάρχει, προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα με τα συστήματα καταθέσεων. μπορούμε να επιλύσουμε όλες τις κρίσεις ε, κατά πάσα πιθανότητα με το παρόν πλαίσιο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κλείνουμε λοιπόν και την ακρόαση αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική. Να περάσουμε στον επόμενο υποψήφιο. welcome uh, Mr. Mauro Grande. He is a counsel to the ECB Executive. Να καλωσορίσω τον κύριο Μάρο Γκράντε, ο οποίο είναι ε, στο εκτελεστικό συμβούλιο. Καλώ ορίσατε στην Επιτροπή μα, στην Επιτροπή Οίκων και συγχαρητήρια για την επίσημη πρότασή σα από την, Ευρωπαϊκή, από την Επιτροπή συγγνώμη, για ε, τη θέση του υπεύθυνου διευθυντή στρατηγικής και συντονισμού στο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξυγένσης. Είχε γίνει ήδη μία ανεπίσημη, άτυπη ανταλλαγή απόψεων, όπως και με τους άλλους υποψηφίους. Και τώρα περνάμε στην επίσημη ακρόαση, η οποία είναι το απαραίτητο στάδιο, πρωτού περάσουμε στην ψηφοφορία, που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα. Και δίνε πάρα αυτά το λόγο στον υποψήφιο για κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις 5 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι θα ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά να συμβάλλω και εγώ στην οικοδόμηση του ε, Συμβουλίου και Μηχανισμού Εξυγίανσης θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα σε μια επαγγελματική σταδιοδρομία που επικεντρώθηκε κυρίω στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ στου ε, πρωταρχικού μου στόχου, εάν διοριστώ σε αυτή τη θέση, για να καταστεί επιτυχής οργανισμό ε, το Συμβούλιο Εξυγίανση. Πρόκειται για έναν ε, θεσμό λοιπόν που θα μπορούσε πράγματι να αλλάξει άρδιν την κατάσταση σε ό,τι αφορά την διαχείριση κρίσεων. Αρχικά, να μείνω στους στόχους ε, τους οποίους ε, θα ήθελα να επιτύχω. Αρχικά θα ήθελα να λειτουργήσει πραγματικά ε, ο μηχανισμός εξυγίανσης ως ενιαίος ευρωνοσιακός μηχανισμός εξυγίανσης. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτονομία των τραπεζών, όμως θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία για να επιτευχθεί και να είναι μάλλον επιτυχής αυτός ο οργανισμός. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ομαλή λειτουργία του συστήματος στο σύνολό του. Δεύτερος στόχος, στον οποίο θα ήθελα να συμβάλλω, είναι η διαμόρφωση μια ισχυρής ευρωπαϊκής ε, προοπτικής. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ενσωματώσουμε όλα τα διασυνοριακά αποτελέσματα μπορεί να έχει η εξυγίανση και σε άλλα στοιχεία του οικονομικού συστήματος και του τραπεζικού κλάδου. Γι' αυτό το στόχο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ε, το ε, Συμβούλιο Εξυγίανσης να έχει και τα απαραίτητα στοιχεία, την απαραίτητη ενημέρωση για να, μπορώ, να μπορεί να αξιολογεί ακριβώς ε, τις ε, είτε ε, του προβλήματος του spillover είτε και για την αξιολόγηση των ε, δημοσίων ε, στόχων κατά την ε, εξυγίανση. Τρίτος βασικός στόχος που θα επιδιώξω είναι η υψηλή ποιότητα εξυγίανσης στο σύνολο του μηχανισμού Ενίας εξυγίανσης. Αυτό θα γίνει και με το Συμβούλιο Εξυγίανσης αλλά και με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Τέλος, θα προσπαθήσω να επιδιώξω ε, μια πολύ ομαλή αλληλεπίδραση και με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο είμαστε υπόλογοι. Και μάλιστα συγκεκριμένα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το SRB μπορεί να ε, εντοπίσει και τα νομικά και θεσμικά προσκόμματα που μας εμποδίζουν ε, να έχουμε αυτή την καλύτερη δυνατή δράση. Γι' αυτό λοιπόν και το SRB και από τη δική του εμπειρία μπορεί να αντλήσει διδάγματα. Ομαλή αλληλεπίδραση επίση θέλω και για, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ξέρετε, έχει και μια διτή ιδιότητα και στο επίπεδο του ανταγωνισμού και στο επίπεδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το Συμβούλιο Εξυγίανση μπορεί να ε, συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον καθορισμό των παγκοσμίων προτύπων εξυγίανση. Αλληλεπίδραση θα πρέπει να υπάρχει και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την εποπτική της ιδιότητα. Πολλές ε, φορές ε, το, Ευρωπα... το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεργάζονται πολύ στενά. Και τέλος, θα ήθελα να διασφαλίσω καλή συνεργασία και με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης εκτός SSM ε, οι αρχές που θα είναι υπεύθυνε ε, για αυτές τις ομάδες ε, εντός του χώρου SSM αλλά και εκτός για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των αρχών εξυγίανσης και διαχείρισης κρίσεων. Ελπίζω πραγματικά να θέσω όλη μου την εμπειρογνωμοσύνη στην υπηρεσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζάλμπα, πρώτος ομιλητής, ευχαριστώ. Πέραν των τεσσάρων στόχων που αναφέρατε, θα ήθελα, αν μπορείτε να μας πείτε, ποιοι είναι οι πλέον σημαντικοί κίνδυνοι και προκλήσεις που ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης και το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης έχουν να αντιμετωπίσουν σε αυτό το νέο στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τι προκλήσεις θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Το πρώτο αφορά το εγχειρίδιο, το rule book το σύνολο κανόνων. Θα πρέπει και εμείς να βασιστούμε στους κανόνες τραπεζικής λειτουργίας. Εμείς βέβαια θα θέλαμε να έχουμε ένα πραγματικό εγχειρίδιο, ένα σύνολο κανόνων, εξυγίανσης πιο συγκεκριμένα, πέρα του τραπεζικού κλάδου. Υπάρχει μια, ένα χαμηλότερο επίπεδο συντονισμού και ευθυγράμμισης εδώ. Γιατί το BRRD, όπως ξέρουμε, μόλις έχει τεθεί σε ισχύ. Δεν το έχουμε ακόμα δοκιμάσει. Μάλλον θα τεθεί σε ισχύ την 1η Πρώτου 2015. Πρέπει λοιπόν από την πράξη να μάθουμε εάν αυτό το σύνολο κανόνων λειτουργεί ορθά στην πράξη. Και πάλι το Συμβούλιο Ξεγίανσης εντοπίζει στοιχεία του συνόλου κανόνων αν εντοπίσει τέτοια στοιχεία που αποτελούν πρόσκομα στην εύρυθμη λειτουργία μα, τότε θα πρέπει να το μεταφέρει αυτό τόσο στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Δεύτερη πρόκληση για μένα. Η εμπειρία σε εθνικό επίπεδο στην εξυγίανση είναι περιορισμένη. Αν συγκρίνουμε την οικοδόμηση του SSM και του SRM, το SSM πράγματι μπορούσε να βασιστεί σε μακρόχρονη εμπειρία των εθνικών αρχών. Δεν μπορούμε το ίδιο με την εξυγίανση, γιατί και πάλι ε, τώρα θεσπίζονται τα, τα συστήματα εξυγίανσης με αφορμή το BRRD και είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να διαμορφώσουμε ταυτόχρονα και την ευρωπαϊκή και την εθνική διάσταση της εξυγίανσης βάσει ενός νέου πλαισίου το οποίο θεσπίζεται και προβλέπεται από το BRRD που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο bailout. Ταυτόχρονα κατά κάποιον τρόπο αυτό το γεγονό ότι τα οικοδομούμε όλα εκ του μηδενό μπορεί να είναι και θετικό. Γιατί μπορεί τελικά στο επίκεντρο του συστήματος να έχουμε μικρότερες αντιστάσεις, να έχουμε ένα ενωσιακό σύστημα. Για να σας πω στην εμπειρία μου ε, για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περάσαμε από διάφορες φάσεις και διάφορα στάδια. έπρεπε να, να υπερπηδήσουμε διάφορα εμπόδια, καχυποψίας, από τις ε, εθνικές ε, κεντρικές τράπεζες. Ήταν δύσκολο να διαμορφώσουμε αυτό το ομαδικό πνεύμα. Ίσως σε αυτή την προσπάθεια τώρα για το SRM να είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο να ξεκινάμε από το μηδέν. Βέβαια, η αξιοπιστία του Συμβουλίου Εξυγίανσης θα βασιστεί και στην ικανότητά του ε, να παράσχει πραγματικά αποδοτική εξυγίανση. Έχουμε διάφορα στοιχεία εδώ. Το βαθμό στον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη διάσωση με ίδια μέσα και ο τρόπος με τον οποίο ε, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα χειριστεί αυτά τα στοιχεία αρμοδιοτήτων που θα του παραχωρηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη μελήτρια η κυρία Μπερέσα από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε υποψήφιε, θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπατε. Συμφωνώ με την ιδέα ότι όταν προσπαθούμε να οικοδομήσουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν αρχίζουμε από το μηδέν, συνήθως τα καταφέρνουμε καλύτερα. Στην περίπτωση όμως αυτή συγκεκριμένα, έχω την εντύπωση ότι Όσον αφορά την αύξηση της ισχύω του μηχανισμού εξυγίανσης, βρισκόμαστε σε ένα deal σχεδόν διακυβερνητικό, που κάθε κράτος μέλος έχει υπερασπιστεί τη δική του ε, εθνική μέθοδο, αντί ε, σε μια ε, ερμηνεία που αντιστοιχεί σε μια οικονομική λογική, γιατί λάβαμε υπόψη βεβαίως τα κριτήρια κινδύνων, αλλά ε, μας υπόθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική φόρμουλα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Η πραγματικότητα της διαπραγμάτευσης ε, του Ταμείου Μετάβασης μήπως αντίκειται ε, τελικά σε, αυτόν τον, σε αυτή την αισιοδοξία σας κατά μιας διακυβερνητικής μεθόδου, κάτι το οποίο δεν ισχύει για το σύστημα εποπτείας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα είναι βασικό καθήκον του Συμβουλίου εντός του συστήματος ε, να γίνει να υπάρξει κάποιο είδους ευρωπαϊκή προοπτική, όπως είπατε. Είναι κάτι το οποίο το Συμβούλιο ε, θα κριθεί μετά από ε, την πάροδο κάποιων ετών και την απόκριση κάποιας εμπειρίας. Πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι ε, το οποίο θα ε, πρέπει ακόμα να το κρίνουμε, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τώρα τη συμφωνία για το Ταμείο Εξυγίανσης που δεν πρέπει να βασίζεται σε ε, διακυβερνητική βάση, όπως είπατε και εσείς θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία θα βοηθούσε παρά το ότι στην πραγματικότητα όντως θα ήταν ε, μια διακυβερνητική μέθοδος ένα εμπόδιο στο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, εγώ παραμένω αισιόδοξο ότι το Συμβούλιο θα καταφέρει να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ε, παρά το γεγονός ότι θα, θα προτιμούσα και εγώ μια άλλη προσέγγιση ίσως ε, να υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία σχεδιασμού τα οποία θα μπορούσαν να ε, τα, τα, μπορούσαμε να τα επιρβούμε μέσω μιας εφαρμογής που θα πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Επερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε βλέποντας και κάνοντας και μαθαίνοντας από τα λάθη μας και στη συνέχεια αυτό το σύστημα μπορεί να καταλήξουμε ότι πρέπει να έχει καλύτερη εξισορρόπηση από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή μετά από το σχεδιασμό ε, με τη διακυβερνητική μέθοδο. Και θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ναι, είναι σημαντικό το Συμβούλιο Εξυγίανση να μπορέσει να τονίζει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους σημαντικούς παίκτε όλα αυτά τα στοιχεία σχεδιασμού τα οποία τελικά αποτελούν ένα σημαντικό πρόσκομα στην πραγματική εφαρμογή, στην αποτελεσματική εφαρμογή. Μία πτυχή σημαντική είναι η διαδικασία λήψη αποφάσεων, την οποία, όπως γνωρίζετε, η οποία, όπως γνωρίζετε, ε, προβλέπει τη συμμετοχή διαφόρων εμπλεκομένων φορέων και ουσιαστικά Υπάρχει δυνατότητα ε, απόρριψης ε, από το Συμβούλιο, από την Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο. Θα δούμε δηλαδή πώς πάει το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος ε, επί της αρχής να πούμε ότι δεν θα λειτουργήσει κάτι. Εμείς θέλουμε το Συμβούλιο Εξυγίανσης να πάρει απόφαση επί πολύ συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή ε, μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό κάτι ε, ή όχι. Απλώς ε, το Συμβούλιο δεν θα προσπαθήσει να αποφύγει την ανάγκη για περισσότερες αλλαγές αν χρειαστεί. Από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές θα ήθελα να παρακαλέσω να μας παρουσιάσετε ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία έως τώρα. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε πάρα πολύ ωραία για τη συνεργασία των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Μιλήσατε λοιπόν πολύ ωραία και εξηγήσατε πάρα πολύ ωραία τι γίνεται για τη συνεργασία μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών. Δεν είπατε όμως τίποτα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή Οίκων. Θα γίνει ασφαλώς ψηφοφορία τη Δευτέρα για το διορισμό σας και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας μιλήσετε για τη συνεργασία σας με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου η απάντηση. Sorry, I, I think I Νομίζω ότι αναφέρθηκα ότι είναι πολύ σημαντική η σχέση με την Επιτροπή σας σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Από δύο πλευρές. Καταρχάς η υποχρέωση λογοδοσίας, γιατί πρέπει να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται και ιδιαίτερος προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά δεύτερον, και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε διαφανείς και προς τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η δεύτερη ψυχή τώρα της συνεργασίας ο βαθμός στον οποίο το Συμβούλιο εντοπίζει εμπόδια που σχετίζονται με τον κανονισμό και την νομοθεσία. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει και το συμφέρει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τα εμπόδια αυτά προκειμένου να αλλάζει η κατάσταση αυτή η τρίτη πτυχή. Περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στο σύνολο του κλάδου για την εξυγένση των τραπεζών, γιατί εδώ το θέμα λογοδοσίας ε, των κρατών μελών που συμμετέχουν στις δικασίες αυτές προς την επικρατεία τους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταστούμε σημαντικός φορέας το παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτό είναι εγγενέ στοιχεία του Συμβουλίου και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είμαστε διαφανείς και να δίνουμε λόγο στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Χούμπνερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, έγινε μία συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ για ένα συμβιβασμό για την ε, εισφορά των τραπεζών τη συμβόλη των τραπεζών σε αυτόν τον ενιαίο ταμείο εξυγίανση. Υπάρχουν κάποιε καινούργιε ιδέε, έχει ακουστεί και η ιδέα κατάργηση του κατοφλίου για τις πληρωμές δεσμεύσεων και μετά το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει από αυτόν. Το ερώτημα μου λοιπόν το εξή. Ποια είναι η άποψή σα για το θέμα αυτό για το πρόβλημα αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχει καταστεί μεγάλο πρόβλημα τελικά το ζήτημα αυτό προκειμένου να λεφτεί μια απόφαση για το 2015, το 2016. Η απάντηση γενικά για τα γενικά, τα βασικά στοιχεία του κανονισμού, του πλαισίου για την ε, συμβολή των τραπεζών. Συμφωνώ με τη βασική ιδέα. Ιδιαίτερα με την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει αρχή αναλογικότητας η οποία να εφαρμόζεται. οι μικρές τράπεζες που θα ωφελούνται λιγότερο από το Ταμείο Εξυγίανσης να συνεισφέρουν λιγότερα. Συμφωνώ και με τη γενική ιδέα ότι οι τράπεζες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερη επικινδυνότητα και θα ωφεληθούν πιο πολύ θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο. Είμαι υπέρ της δομής αυτής λοιπόν. Για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρατε, για να είμαι ειλικρινής δεν έχω κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δεν είναι ένα θέμα δεν έχω κάποια προσωπική τοποθέτηση. Δεν προτιμώ να μην σας, ε, να σας το ομολογήσω αυτό παρά να σας ε, υποστηρίξω γενικότητες. Η διαφορά μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών, δεσμεύσεων πληρωμών έχει να κάνει με οποιοδήποτε είδος ταμείου. Αυτό το αναφέρουμε και σε διάφορα το του το Loss absorbing capacity στο παγκόσμιο προσκήνιο. Υπό ένα σημείο, μοναδικό σημείο εισόδου, η... το επίπεδο TLAC θα πρέπει να κατανέμεται σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσω των ισολογισμών ή μέσω εγγυήσεων από το κεντρικό σημείο της επιχείρησης. Αν υπάρχει εγγύηση, φυσικά δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχουν τα χρήματα όταν θα τα χρειαστούμε. Ενώ η πληρωμή σε ρευστό εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Δεν είμαι μετακινητός εκ πρώτης όψεως θα έλεγα ότι κλείνω μάλλον στο να υπάρχει πληρωμή σε είδος, προκειμένου να υπάρχει ρευστότητα, αν χρειαστεί. Γιατί όταν κληθούν οι τράπεζες ε, να πληρώσουν την ώρα που θα παραστεί η ανάγκη, θα υπάρχει πάλι το θέμα της προκυκλικότητας και ενδεχομένως τα πράγματα να δυσκολεύσουν. Τέτοιου είδους σκέψεις έχω στο μυαλό μου και πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη που με οδηγούν σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι καλύτερα να υπάρχει ρευστότητα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι πιο ακριβής. Δεν έχω κάποια αμετακίνητη άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κανείς άλλος? Στη διαδικασία Catch the Eye, αν όχι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ την ακρόαση. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Η ψηφοφορία, όπω ξέρετε, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. try to anticipate a little bit also the hearing. Προσπαθούμε. Θα περιμένουμε λίγο τον κύριο Λατινιέμι. Καταφθάνει όπου να είναι. Παρακαλώ, μείνετε στην αίθουσα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών. How long? Oh, I was on the stairs, so even less. Yes. Waiting instruction from the secretariat. Whether. Αναμένουμε οδηγίες από τη γραμματεία, λέει ο Πρόεδρος. Whether some speakers of political groups are coming, in this case we wait. Κατά πόσο έρχονται εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, αν ναι, να τους περιμένουμε. We can start. Great. Welcome. Καλώς ήρθατε, ε, κύριε Τίμο Λοϊτινιέμι. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Ε, είστε διευθυντής ε, του Κρατικού Ταμείου Συνταξιοδότησης. Είχατε μία πρώτη ενταλλαγή απόψεων με την ομάδα εργασίας για την Τραπεζική Ένωση της Επιτροπής μας. Ε, τώρα έχετε επιλεγεί επισήμως ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας αυτή. Και τώρα θα γίνει αυτή η επίσημη ακρόαση, η οποία μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Και θα, ε, αρχίσουμε με τα εισαγωγικά σας σχόλια για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου για τα καθήκοντα αντιπροέδρου του ε, Συμβουλίου Εξυγίανσης, αλλά και για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Καταρχάς θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και μετά θα μπω στα συγκεκριμένα καθήκοντα του αντιπροέδρου ε, στο ε, ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Είναι ένα σημαντικό τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης. Το 2008 ήταν ένα σημείο ή ε, ήταν ανεπαρκής ε, η η δράση μας ε, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και το τίμημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και για τις τράπεζες και για την κοινωνία ολόκληρη. Τα, οι εκτιμήσεις κόστους μόνο για τις Ηνωμένε Πολιτείες ήταν πάνω από 43 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρώπη επίσης ε, επλήγει ε, το κυβερνητικό χρέος ε, εν μέρη το φέρει ο οικονομικός τομέας, όμως πρέπει η Τραπεζική Ένωση να αναλάβει δράση επιγόντως. Ε, ο ενίος μηχανισμός εξυγίανσης και το Συμβούλιο ε, σκοπό έχει να ε, βοηθήσει το, την οικονομία, να αντιμετωπίσει τις, ε, τα προβλήματα. Είναι ε, ένας συντονιστικός φορέας ε, για την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών φορέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν κανόνες συγκεκριμένοι, στους οποίους συμμετείχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφώνως με τις, τα απορίσματα του συστήματος οικονομικής σταθερότητας και του G20. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τον ενιαίο νέο μηχανισμό εξυγένση που για μένα είναι βασική καινοτομία στο νέο ε, μηχανισμό για τα ε, προβληματικά ε, τραπεζικά ιδρύματα όπως είναι το bail-in γιατί το bail-out θα υποκατασταθεί από ένα νέο μηχανισμό που είναι το bail-in. Στο bail-in το χρέος εκτός των κυβερνητικών καταθέσεων και άλλων προκαθορισμένων υποχρεώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές περιπτώσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι μια καινοτομία και χρησιμοποιείται ως μια φαιά ζώνη ώστε να μην πλήττονται οι φορολογούμενοι από τον ενδεχόμενο αντίκτυπο μιας διάσωση. Έχει οδηγήσει εν μέρη τι τράπεζε ε, στην ύπαρξη, στη δημιουργία μέσων που μπορούν να του βοηθήσουν από απορροφήσουν ε, το ε, σοκ ε, μιας τέτοιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα μεγάλα αυτά πλήγματα, τα χρηματοπιστωτικά, μπορούν να προκύψουν από διάφορες πλευρές. Είναι κάτι το οποίο έχει αξιολογηθεί στην επισκόπηση των, ε, ε, του ποιοτικού ενεργητικού. Υπάρχουν κάποια σενάρια, ε, κάποια χειρότερα σενάρια, τα οποία ε, σκιαγραφήθηκαν, κάτι το οποίο εκτίμησε όλο ιδιαι, όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας και υπήρξε, υπάρχουν πλέον αρκετά μέσα και αρκετό κίνητρο ώστε να ενισχυθούν ε, οι δομές ήδη και το 2014. Να περάσω τώρα στο ρόλο του Αντιπροέδρου στον, το Συμβούλιο Εξυγίανσης. Ε, αυτά τα καθήκοντα ε, είναι Τριπλά ε, είναι το Ταμείο Εξυγίανση, η συμμετοχή ε, στα καθήκοντα της εξυγίανση όπως θα αποφασίσει το Συμβούλιο και θα συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και θα είναι υπεύθυνο για τις ε, εταιρικέ υπηρεσίες. Θα καλύψω αυτές τις τρει ιδιότητες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το Διευθυντήριο για το Ταμείο Εξυγίανσης. Να δούμε δηλαδή πόσες καταθέσεις, το ποσό των καταθέσεων που ε, καλύπτεται. 55 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε 8 ε, χρόνια από τις αρχές του 2016 ελπίζουμε για το Ταμείο Εξυγίανσης πριν υπάρξει, πριν συγκεντρωθεί αυτό το ποσό θα υπάρξει ένα σύνολο κανόνων που θα είναι απαραίτητα θα πρέπει να, γίνουν, να γίνει η ρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι οι πολιτικές επενδυτικές έχουν πάντοτε σχέση με ένα συγκεκριμένο σκοπό και πρέπει να διαμορφωθούν πριν αρχίσει να ισχύει το Ταμείο. Ε, ε, δρομολόγησε ένα λεπτομερέ σχέδιο η Επιτροπή εδώ και δύο εβδομάδε. Ο στόχο του συστήματο ε, των τυσίων εισφορών στο Ταμείο είναι δίκαιο και εξισορροπημένο βάσει του προφίλ κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεύτερον, ο πρόεδρος ε, ενεργεί ε, ως μέλος του Συμβουλίου στις ε, διαδικασίες εξυγίανσης όταν άλλες μέθοδοι ε, για την ενίσχυση των τραπεζών είναι ανεπαρκείς και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο καθιστά τις τράπεζες ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται πάντοτε για μια διαδικασία εξισορρόπησης, καλύτερος ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών, όπως επίσης και στέρεα βάση για την ανάπτυξη των θέσεων απασχόληση και τη ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Αντιπρόεδρο είναι υπεύθυνο για τις εταιρικέ υπηρεσίες, κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά θέματα, από ανθρώπινο δυναμικό μέχρι διαχείριση, θέματα διαχείρισης και θέματα ε, τεχνολογίας των πληροφοριών. Ε, το, τα καθήκοντα του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το καθήκον του Προέδρου επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση του Ταμείου Εξυγένσης που είναι πραγματικά ένα μοναδικό καθήκον. Εγώ θα ήθελα να συμμετέχω στην ενίσχυση στεναρών χρηματοοικονομικών συστημάτων ώστε να μπορέσουμε ε, να έχουμε μακροπρόθεσμες προοπτικές ευημερίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να ακούσω ερωτήσει από τα μέλη τη επιτροπή σα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ομιλητή από πλευρά ΕΛΚ, ο κύριο Παύλο Ζάλμπα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, κύριε υποψήφιε, για την ε, ομιλία σας. Μιλήσατε για τους Ευρωπαίους ε, πολιτές. Ελπίζουμε πραγματικά αυτό να αποβεί σε όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. επί τη ευκαιρία και εφόσον αναφερθήκατε και, για και στη δημοκρατική λογοδοσία, πώς σκοπεύετε ακριβώς να εφαρμόσετε αυτή την αρχή της ε, δημοκρατικής λογοδοσίας ό,τι αφορά τον μηχανισμό ε, εξυγίανσης και πώς προτίθεστε να συνεργαστείτε με το Κοινοβουλίο μας. Σας ευχαριστώ. Συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου Επιτροπής και SRM είναι εξαιρετικά σημαντική. Το Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει αυτόν τον κανονισμό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, να λειτουργεί σωστά αυτή η συνεργασία. Κατανοώ ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ακριβώς ε, για να λειτουργήσουν ως ασφαλιστικές δικλείδες για τη συνεργασία μεταξύ ε, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και του Συμβουλίου Εξυγίανσης. Πραγματικά λοιπόν πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές θα υποφεληθούν αυτής της συνεργασίας και είναι κάτι το οποίο μας αφορά ιδιαίτερω, μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Η κυρία Μπεχάη από πλευρά Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε υποψήφια, για τη θέση του Πρόεδρου. Σα ευχαριστώ που περιγράψετε πολύ ωραία πώ βλέπετε κι εσεί τον ειδικό σα ρόλο. Θεωρώ ότι το βήμα που κάνουμε με τη θέσπιση αυτού του ταμείου είναι πολύ σημαντικό. Έχω όμως ένα σημείο προβληματισμού που συνδέεται με τον διακυβερνητικό χαρακτήρα ε, που έχει πάρει όχι η πλευρά της εποπτείας, που είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται λογικό και ότι πρέπει να κινηθεί προς την ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, η χρηματοδότηση του Ταμείου Εξεγίανσης έχει λάβει διακυβερνητική διάσταση. Μήπως θεωρείτε ότι αυτό θα μεταφερθεί και θα μεταφραστεί σε εντάσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και ότι θα έχουμε δυσκολίες θα έχετε μάλλον δυσκολίες να ασκήσετε με αντικειμενικό τρόπο ε, την ιδιότητά σας, τα καθήκοντά σας στην εξυγίανση. Και σε ό,τι αφορά τη σύνθεση ε, των ε, ταμείων εξυγίανση, θα ήθελα να σχολιάσετε πιο συγκεκριμένα. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο τρόπος χρηματοδότησης διασφαλίζει κατά τη διάρκεια τη μεταβιβητική περίοδου εννοώ τώρα διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία των μελών ε, του Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένη και τη σύνθεσή του. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η χρηματοδότηση του Ταμείου Εξυγένσης σε ένα βαθμό έχει αποφασιστεί σε ένα βαθμό και τα υπόλοιπα θα αποφασιστούν στην πορεία. Θα είναι λοιπόν χρηματοδότηση εξάντε. Εν μέρη θα υπάρχει καταποκοπή εισφορά και εν μέρη θα βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Μετά θα έχουμε σε ε, δεύτερο βαθμό και εξπόστε εισφορές, αν αυτό καταστεί απαραίτητο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μετά υπάρχουν και άλλες δύο δυνατότητες αν υπάρχουν ε, καταστάσεις επίγουσης ανάγκης, ο δανεισμός από άλλες αρχές και άλλους μηχανισμούς εξυγίανσης και τέλος υπάρχει και η δυνατότητα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Για το πρώτο τμήμα των εισφορών εξάντε. Όπως είπατε, μπορεί να υπάρξουν διακυβερνητικές εντάσεις, αλλά από ό,τι βλέπω, ο κανονισμός είναι, έχει συνταχθεί, είναι σαφέστατος ότι ο στόχος του Ταμείου είναι πολύ σαφής και το επίπεδο στόχος της χρηματοδότησης είναι σαφής. Και 55 δις ευρώ στο σύνολο. Είναι ένα ποσό που νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί επαρκέ ε, για να καλύψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω η διαδικασία να είναι ε, ομαλή, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και συζητήσει ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χούμπνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει πολύ κατακριματισμό στον τραπεζικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί θα έχετε κυρίως τράπεζες που έχουν μεγάλη εμπειρία σε διασυνοριακή δράση. για τράπεζες εξυγίανση που συμμετέχουν σε διάφορα μέρη. Πώς αντιμετωπίζετε την πρόκληση των εσωτερικών ζητημάτων. Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερες ε, συνθήκες σε ό,τι αφορά την εξυγίανση, τη διασυνοριακή και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά, ιδιαίτερα σε διάφορα αφορά τράπεζες που δρούν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τη Ευρωζώνης. Τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης και τα πρώτα βήματα γίνονται με τη σύσταση του Συμβουλίου. Τα διασυνοριακά καθήκοντα είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση λόγω του νομικού καθεστώτος σε διάφορες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς βρίσκεται στη φάση της διαδικασίας αντιμετώπισης των διασυνοριακών προβλημάτων. Μακροπρόθεσμα, ασφαλώς, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της Ευρωζώνης, των ευρωπαϊκών χωρών και των λοιπόν ε, ιδρυμάτων. Τέτοιου είδους συνεργασία είναι απαραίτητη στο επίπεδο του G20 σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πρόκειται για τις βασικές δυνάμεις για την προώθηση των ζητημάτων αυτών και το Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει την ιδιότητα και την ευθύνη συντονισμού με άλλες ε, αρχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρος. Κανένα άλλο σχόλιο, καμία άλλη παρατήρηση. οποία ωστόσο ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, συντομότατη αυτή ακρόαση, η οποία ωστόσο ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη και χρήσιμη και απαραίτητη και επίσης θετική. Ανυπομονούμε λοιπόν ε, και προσβλέπουμε στην ψηφοφορία η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς και τους υπόλοιπους υποψηφίους για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τις προηγούμενες επαφές που είχαμε. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία καθ' όλη τη διαδικασία αυτή και προσβλέπουμε στην θετική ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής προκειμένου να υπάρξει τελικά το Συμβουλίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξυγίανσης. Πολύ βασικό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον υποψήφιο αντιπρόεδρο, λέει ο πρόεδρος.